Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Βρισκόμαστε σε ένα νέο περιβάλλον, μια από τις παλιές αίθουσες συνεδριάσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορούμε λοιπόν σήμερα να ξεκινήσουμε, αλλά λόγω της ημέρας για πολλούς από εμά, όπως μπορώ να διαπιστώσω, είναι μια μέρα που έχουν πολλοί από εμά άλλες υποχρεώσεις, αλλά βλέπω ότι έχει βελτιωθεί το ηθικό σας με την ε, ε Τυρκουάς και έχουμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε με το πρόγραμμα μας για σήμερα με μεγαλύτερο ενθουσιασμό. Λοιπόν, το πρώτο σημείο είναι η έγκριση της διάταξης. Αν δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχει εγκριθεί. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Να σας πω τα εξής. Την, την προπροηγούμενη εβδομάδα πήγε μια αντιπροσωπή από εμάς στην συνδιάσκεψη του ΟΗΕ για την ε, βιοποικιλότητα Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι υπήρξε στο τέλος κάποια συμφωνία και η διαδικασία του ΟΗΕ δεν έχει εξοκύλει τελείς, αλλά χάρη στην συνδιάσκεψη στην Αγκόγια έχει προχωρήσει λοιπόν. Τουλάχιστον υπάρχει ένα αποτέλεσμα το οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι ικανοποιητικό από την Αγκόγια. Ε, γνωρίζετε ότι έγιναν οι εκλογές στην ε, Βουλή των Αντιπροσώπων και την Γερουσία. Το που έχετε παρακολουθήσει αυτό, ξέρετε τι σημαίνει αυτό για την ε, κλιματική αλλαγή εν ώψη και της συνδιάσκεψης της Κανκούν. Τα πράγματα δεν γίνονται ευκολότερα λοιπόν και θα πρέπει να δούμε αν τα δύο μεγάλα κόμματα στην Αμερική θα μπορέσουν να έχουν μια πιο λογική στάση και να μπορέσουν να προετοιμαστούν για μια συμφωνία για τα κλιματικά θέματα που να είναι πιο ευνοϊκή. Επίσης, λάβαμε πρόσφατα μια ανακοίνωση της Κομισιόν σε σχέση με το πρωτοκόλλο του Κιώτο και σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει λόγω αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση <coughs> το 8% μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. 10,4 είναι αυτό το οποίο έχουν επιτύχει τα 15 κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα παλιά, και 14,3 στο σύνολο των 27 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεπερνούμε λοιπόν το 8% βέβαια είναι σαφές ότι βοήθησε η οικονομική κρίση άκοντες όλοι να μειώσουμε τις εκπομπές μας σε επίπεδο διοξιδίου του άνθρακος. Αλλά τουλάχιστον είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επιτύχει το στόχο του 8% ο είχε τεθεί. Επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στις 14 και 15 μέχρι τις 15 θα παρουσιαστεί μια ταινία από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Άγρια Πανίδα και τη Φύση για τον Τόνο. Όποιος θέλει λοιπόν και όποιος ενδιαφέρεται για την αλία και τα θέματα αυτά της διατήρησης των αλλιευτικών αποθεμάτων μπορεί να έρθει σε αυτή την αίθουσα στις 14 και 15 να δει αυτή την ταινία. <clears throat> Αυτό λοιπόν για τις ανακοινώσεις που ήθελα να σας δώσω. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 3 της ημέρησης διάταξης. Ενίσχυση της χημικής, βιολογικής, ραδιολογικής και πυρηνικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. ΧΒΡΟΠ είναι το σχέδιο δράσης. Η Κατίκα Λέοτάτ είναι η συγγήτρια για το ζήτημα αυτό. Και έχουμε και μία σειρά τροπολογιών οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν έχετε φέρει όλη την ε, κάρτα ψηφοφορία σας. Εγώ τουλάχιστον τη δική μου την έχω φέρει. Στην περίπτωση που δεν θα έχουμε σαφείς πλειοψηφίες θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και ξεκινούμε με την ψηφοφορία. 7 και 8 από κοινού ψηφίσουμε. Ψήφι υπέρ. 7 και 8. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές γίνονται δεκτές. Τροπολογία 9. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 11 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 12 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 14. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για τη 14. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, μια στιγμή. Δεν λειτουργεί το μηχάνημά σας. Δεν λειτουργεί, δεν λειτουργεί. Πάρτε το διπλανό μηχάνημα. Ναι. Επαναλαμβάνουμε γιατί η κυρία Τζουαρντίνη είχε πρόβλημα με το μηχάνημα Τσούτη και αυτό δουλεύει. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε για τροπολογία 14. Πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 20 κατά. Γίνεται δεκτή η τροπολογία 14. Πηγαίνουμε στην 15. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά απόχες δεκτή 20 ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 υπέρ κατά αποχές δεκτή 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 σε δύο τμήματα πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται το πρώτο τμήμα. Δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Πάει και αυτό. Απορρίπτεται. 27. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αιτιολογικές σκέψεις. Υπαριθμόν 1. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. 2 ψήφι <clears throat> κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές επίσης δεχτή. Τελική ψηφοφορία λοιπόν, ηλεκτρονικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 48 ψήφοι υπέρ, ομόφωνα, καμία ψηφός κατά καμία Αποχή συγχαρητήρια κυρία Λεωτάρτ. Περνάμε λοιπόν στο σημείο 4. Ευρωπαϊκή οικονομική λογαριασμή. Μία έκθεση την οποία μου έχουν ε, εμπιστευτεί σε μένα τον ίδιο οι συντονιστές. Και έχουμε εδώ μια σειρά τροπολογιών, μια μακρά σειρά τροπολογιών που πρέπει να ψηφίσουμε. Τροπολογία 6. Ψήφι ΠΕΡ Κατά. Αποχές δεκτή. 12 της Οικονομικής Επιτροπής. οικονομική 12. Ψήφι ΠΕΡ Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Οικονομική 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Πέρας φοφορίες. 26 υπέρ, 23 κατά. Δεκτή. 7 ψήφι υπέρ. κατά αποχές δεκτή 29 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27. Υπάρχουν 27. Οι προηγούμενες έχουν εκπέσει. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9. Ψήφι υπέρ. κατά αποχές δεκτή. Yeah. Äh, 15 της Οικονομικής Επιτροπής, ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 Κρίστα Κλάς. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 9. Το δεύτερο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33. Υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 <clears throat> υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή 36 υπέρ κατά αποχές δεκτή οικονομική 16 ψήφι υπέρ κατά αποχές δεκτή 37 υπέρ κατά αποχές δεκτή Οικονομική 17. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Γιατί είναι 38. Ψηφίσατε όλοι πέρα ψηφοφορία. Δεκτή με 27 ψήφους υπέρ 21 κατά, 39 ψήφοι υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 11 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 12 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 14 ψήφι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Οικονομική 19. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 43. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 44. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 45. Ψήφι υπέρ. Κατά. Απόχες. Δεκτή. 46 ψήφι πέρα. κατά αποχές δεκτή οικονομική 20 ψήφι πέρα κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 48 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή αιτιολογικές σκέψεις οικονομική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οικονομική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Οικονομική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Απορρίπτεται. Οικονομική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Αλλά μπορούμε να ελέγξουμε ίσως. Οικονομική 4 κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. <clears throat> Πέρας ψηφοφορίας πράγματι εγκρίνεται. Τροπολογία 1 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Οικονομική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο για τη 18. περας ψηφοφορίες, ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, πράγματι, σαφώς, 30-18. 19 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Οικονομική 7 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 20 ψήφοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Οικονομική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 3 ψήφοι υπέρ κατά αποχές δεκτή. 4 Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 21. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 22. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ή μάλλον ας κάνουμε έλεγχο για την 24. Πέρας. Εγκρίνεται πράγματι. 25 ψήφι υπέρ. Κατά. Εγώ νομίζω, νομίζω την ίδια πλειοψηφία. Ας κάνουμε όμως και ένα έλεγχο για την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Με την ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Ερχόμαστε στην τελική ψηφοφορία, λοιπόν, ηλεκτρονικά παρακαλώ, αρχιδη ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 39-2 με 6 εποχές και το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Λήξεις. 40 ψήφοι υπέρ, 4 κατά, 4 <coughs> αποχές. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Και ούτως ή άλλως Αυτό το θέμα θα είναι ένα ζήτημα το κατά πόσο αυξάνεται το παγκόσμιο περιβαλλοντολογικό κεφάλαιο ή μειώνεται και επομένως θα πρέπει να κάνουμε τις απαραίτητες προσαρμογές στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ερχόμαστε στο σημείο 5 της ε, ημερησίας διάταξης τώρα. Αξιολόγηση διαχείρισης της γρήπης H1N1 κατά τη διάρκεια του 2009 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λεγόμενη γρήπη των χείρων, όπως ονομάστηκε σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Μιχέλ, Μισελ Ριβαζή είναι η συγγήτρια, η οποία θα μας παρουσιάσει την έκθεσή της και της δίνω το λόγο για να μας παρουσιάσει την έκθεσή της. Μισελ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι σε επίπεδο διαχείρισης αυτής της γρήπης α ή τα 1 1 ε, είχαμε ζητήσει μία μελέτη ε, αλλά δυστυχώς ε, η συνδιάσκεψη των Προέδρων ε, αρνήθηκε να οργανώσει αυτή τη ε, μελέτη. Έγιναν όμως κάποιες ακροάσεις. Η μία ακρόαση έγινε εδώ σε αυτή την Επιτροπή και είχαμε τους υπεύθυνου όταν είχε ξεσπάσει η επιδημία και ρωτήσαμε Τι θα έκαναν σε μια τέτοια περίπτωση. Ε, τι διαπιστήσαμε. Ότι όταν ξέσπασε αυτή η επιδημία ή τα ένα νη ένα, τον Μάιο ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η κυρία Τσάν δηλαδή, είχε πει ότι πρόκειται για μια καλοήθη γρήπη. Όμως παρόλα αυτά το Ιούνιο του 2009 ε, ανέβηκε το επίπεδο συναγερμού. Φτάσαμε στο επίπεδο 6. Μετά αρχίσαμε να συζητάμε για τα κριτήρια καθορισμού της πανδημίας. Το 2009 η πανδημία ήταν μια γεωγραφική επιδημία όχι όμως ε, με βάση τον αριθμό των θανάτων. Και αυτό δημιουργούσε προβλήματα, διότι οποιαδήποτε ασθένεια, εάν δούμε πώς εξαπλώνεται γεωγραφικά, αλλά δεν εξατάνσουμε την σοβαρότητά της, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν πανδημία. Από την, άλλη φορά, από την άλλη πλευρά υπήρχαν ε, τεράστια έξοδα ε, για την αγορά των ε, εμβολίων. Δισεκατομμύρια δαπανήθηκαν στην Γαλλία, 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ για να αγοράσουμε εκατομμύρια εμβόλια. Και μονάχα 8 εκατομμύρια χρησιμοποίησαμε. Μετά είχαμε το πρόβλημα της στρατηγικής εμβολιασμού δεν υπήρχε ένα συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Υπήρχαν διαφορές κράτη-μέλη θεώρησαν ότι έπρεπε να γίνει μια στοχοθετημένη, στοχοθετημένος ε, εμβολιασμό, δηλαδή τα παιδιά, οι έγκοι, τα οι, άτο... οι διαβητικοί, οι νεφροπαθείς και άλλοι που και άλλα κράτη που θέλουν να κάνουν ένα μαζικό εμβολιασμό. Επομένως, σε θέματα συστάσεων θα πρέπει να δούμε και ποιος, ποια ήταν η αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού και μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ξέρετε ότι η Ευρώπη έχει ένα πιο συντονισμένο όραμα Εξού και θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα τι είδου εμβολιασμό χρειάζεται να κάνουμε. Μετά είχαμε διάφορες ακροάσεις και είχαμε οργανώσει και μία ακρόαση για την δεοντολογία των εμπειρογνωμόνων και τη σύγκρουση συμφερόντων και την διαφάνεια θα πρέπει να βελτιώσουμε την διαφάνεια και την πρόσβαση στην βιβλιογραφία, στα έγγραφα. Ο Ευρωπαϊκός ε, Διαμεσολαβητής για τον οργανισμό φαρμα, Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ε, λέει ότι ε, οι μελέτες που γίνονται για την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και την τοξικότητα των φαρμάκων θα πρέπει να είναι προσβάσιμες στο κοινό, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει τώρα. Επίσης, την, η ευθύνη για τις παρενέργειες ε, ε, των εμβολίων. Ποιος είναι υπεύθυνο, διότι δεν ήταν τα, οι, οι φαρμακευτικές εταιρείες, ε, τα, φαρμακευτικά εργαστήρια τα οποία ήταν υπεύθυνα για τις παρενέργειες, αλλά τα κράτη-μέλη ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως, θα πρέπει σε περίπτωση εμβολίων, οπωσδήποτε, τα φαρμακευτικά εργαστήρια να είναι υπεύθυνα για τις παρενέργειες. Επίσης, χρειαζόμαστε περισσότερη ανεξαρτησία έχουμε δύο υπηρεσίες πάρα πολύ σημαντικές στην Ευρώπη που είναι το κέντρο ελέγχου των μολυσματικών νόσων και έχει σαν στόχο να αξιολογεί τους κινδύνους και μετά έχουμε και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Θα πρέπει οπωσδήποτε αυτοί οι δύο οργανισμοί, κυρίως ε, το Κέντρο για τον Έλεγχο των Μολυσματικών Νόσων, να ε, εξετάζει το κατά πόσον και εμείς όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ε, ε, αναφέρει μία πανδημία θα πρέπει να δούμε κατά πόσον εμείς έχουμε τα ίδια κριτήρια. Δηλαδή κάθε ε, οργανισμός θα πρέπει να έχει να αναλαμβάνει κάποια ευθύνη. Επίση, θα πρέπει να έχουμε και κάποια ευελιξία όσον αφορά τα επιστημονικά δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μα. Εάν δούμε ότι η γρήπη δεν είναι τόσο σοβαρή όπω πίστευαν αρχικά οι εμπειρογνώμονε, θα πρέπει να κάνουμε μια νέα ε, ε, αξιολόγηση της στρατηγικής μας. Κάτι τέτοιο δεν έγινε εδώ. Το 2010, το 2000, τον Ιούλιο του 2010 λήξαμε το συναγερμό της πανδημίας, που δεν υπήρχε πλέον καμία επιδημία σε κανένα κράτος μέλος, άρα χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία. Δεύτερον, θα πρέπει αυτό το, κέντρο, Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη και τον Έλεγχο των, των Ασθενειών να ε, έχει ένα, μια δικά, δικιά του κλίμακα συναγερμού ανεξάρτητη από τους άλλους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται μια σωστή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των εμβολιασμών. Έγιναν πάρα πολλέ ακροάσεις εμπειρογνωμόνων που έδειξαν ότι υπάρχει μια συνήθεια να εμβολιάζουμε. Αλλά είναι αποτελεσματικός ο εμβολιασμός. Εκεί δεν ξέρουμε. Άρα πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνονται περισσότερε αξιολογήσει όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών. Επίση, πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ε, έγκριση που δίνουμε για τις ε, ε, πιο επιταχυμένες διαδικασίε. Λοιπόν, έννοια διαφάνεια τώρα θα πρέπει να γίνει μια ακρόαση ε, για την αποτελεσματικότητα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, για, την, ε, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον έλεγχο και την ε, τον έλεγχο και την διάδοση των ασθενειών και θα πρέπει να γίνονται, να έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια και για τις κλινικές δοκιμές και για τις παρενέργειες των φαρμάκων και επίσης, και, κάτι, και εδώ υπήρξε κάποια πρόοδος, διότι στα διάφορα κράτη-μέλη εμφανίστηκαν διάφορα σκάνδαλα, θα πρέπει να προσέξουμε τη σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει να να υπάρχει μια εμπιστοσύνη προς τους εμπειρογνώμονες που χρησιμοποιούμε. Ο Ευρωπαίος πολίτης πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους. Επομένως, θα πρέπει να μπορούμε να έχουμε δημόσιο έλεγχο αν θέλετε. Ε, δηλαδή ένας εμπειρογνώμονας μπορεί να πει εγώ είμαι ανεξάρτητος, δεν εργάζομαι για κανένα εργαστήριο. Αυτό όμω μπορεί να μην συμβαίνει. Άρα θα πρέπει κάποιο να τον ελέγχει αυτόν τον άνθρωπο. Πρέπει να υπάρχει ένα οργανισμό ελέγχου. Επίση ε, θα πρέπει και οι, οι, οι, οι ψηλόβαθμοι ε, δημόσιοι υπάλληλοι να, και οι ψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να ελέγχονται με κάποιο τρόπο. Επίσης, όσον αφορά τη συνεργασία, η τελευταία ακρόαση που έγινε τον Ιανουάριο που θα γίνει μάλλον τον Ιανουάριο και σας προσκαλώ σε αυτήν, ε, θα έχει σαν στόχο τη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη. Άρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να ορίσουμε τον ρόλο της, αρμόδιας, της αρμοδιότητας και τις ευθύνε και της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Διάδοση των Ασθενειών και των κρατών μελών. Επομένως θα πρέπει να έχουμε μια διαδικασία που θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αγοράζουν μαζικά τα φάρμακα. Θυμόσαστε ότι όταν είχαμε εκείνη την επιδημία υπήρχαν κράτη τα οποία δεν είχαν τα οικονομικά μέσα να αγοράσουν το εμβόλιο. Εάν όντως ο ιός αυτός ήταν θανατηφόρος, τι θα γινόταν. Τα, η Γαλλία, η Αγγλία θα, μπορούν, θα είχαν τα χρήματα να αγοράσουν τα εμβόλια, τα, τα άλλα κράτη-μέλη όμως όχι. Άρα θα πρέπει να έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε μαζικές αγορές. Από τη στιγμή όμως που είμαστε σίγουροι ότι ο εμβολιασμό αξίζει τον κόπο. Είναι σωστή η, η σχέση ωφέλους και κινδύνου. Ένας, μια άλλη πτυχή, την οποία πρέπει να προσέξουμε, είναι η χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια σαφή εικόνα για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών. Για, τον Ευρωπαϊκό, για, το, για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διάδοση των Ασθενειών δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, διότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί άμεσα. Άρα εκεί μπορούμε να βλέπουμε. Όμως, ε, για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, το 80% της χρηματοδότησης προέρχεται από τις, από τα φαρμακευτικές εταιρείε. Και αυτό σας το λέω γιατί, ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανεξάρτητη και θα πρέπει να αυξήσουμε την αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη των πολιτών μας απέναντι σε αυτούς του οργανισμού. σε αυτούς οργανισμούς. Άρα, θα πρέπει να δράσουμε αποτελεσματικά, γιατί βλέπουμε ότι μετά την τελευταία κρίση υπάρχουν πολύ λιγότερα άτομα τα οποία θα ήθελαν να εμβολιαστούν για κάποια άλλη νόσο. Γιατί είδανε τι, τι έγινε το φιάσκο με την, ε, με την προηγούμενη επιχείρηση. Άρα θα πρέπει να βρούμε τρόπους να ανορθώσουμε την εμπιστοσύνη ανάμεσα σε όλους τους ε, ενδιαφερομένους ε, φορείς. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, Ριβαζή για την έκθεσή σας για την διαχείριση της γρήπης ΙΤΑ1-1. Υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να παρέμβουν. Υπάρχει στις 11 ώρα πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε τον πρέσβευτή της Χιλής, μετά έχουμε την καταστροφή στην Ουγγαρία. Στην Ουγγαρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Καταρχήν να υπογραμμίσω τη σημασία αυτής της έκθεσης που είναι έκθεση πρωτοβουλία, αλλά σημαντική διότι αγγίζει θέματα τα οποία είναι ουσιώδη βασικά. Καταρχήν είμαστε σε θέση σήμερα να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία. Το συστήμα που υπάρχει ε, για να αντιδράσει κανείς είναι το κατάλληλο για να τα τους κινδύνους που υπάρχουν ε, με την εμπειρία του παρελθόντος βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπάθησε να εφαρμόσει κάποιο σύστημα για την αντιμετώπιση μολυσματικών νόσων και ένα σύστημα συναγερμού για να μπορέσει να παρακολουθήσει κανείς μολυσματικές νόσεις. Υπάρχει και επιτροπή για όσον αφορά την ασφάλεια εναντί τέτοιων νόσων, αλλά το θέμα είναι όλα αυτά αρκούν για να αντιμετωπίσουμε μια πανδημία. Φυσικά, ε, σε αυτά τα θέματα βλέπουμε πώς αντιέδρασε κάθε χώρα μέλος και λογικά σε μια ε, απειλή που το να υπάρχει. Και υπήρχε μια βεβαιότητα όσον αφορά αυτή την απειλή. Είδαμε όμως η αντιδράση ήταν ε, ε μονομερής χωρίς κάποια συλλογικότητα. Υπάρχει το θέμα της συνεκτικότητας σε αυτή την αντίδραση, αντιδράση που υπήρχε σε ένα συντονισμό ανάμεσα στις κράτες μέλη ε, για να μπορέσει κανείς να ενημερώσει όσον αφορά τον ιό πανδημίες και φυσικά η απάντηση μπορεί να δώσει κανεί ότι δεν είμαστε έτοιμοι σήμερα να αντιμετωπίσουμε με τον καταλληλότερο τρόπο σε ένα τέτοιο πρόβλημα. Και οι ίδιες χώρες έφτασαν αυτό το θέμα ε, το 12 Οκτώβρη 2010 όταν έγινε το Συμβούλιο όπου είπαν ότι είναι αποφασισμένες οι χώρες μέλη να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα ε, για να αντιμετωπίσουν τέτοιους κινδύνους. Έχουμε μια, λοιπόν μια ευκαιρία και θα πρέπει να ενισχύσουμε το συντονισμό, τη συνεργασία όσον αφορά σε θέματα υγιεινής ανάμεσα στις χώρες μέλη για να διασφαλίσουμε, να προστατεύσουμε τον πολίτη και να υπάρχει μια πρόσβαση ε, στην ε, αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων σε όλους. Ε, χαιρετίζω την ε, εισηγήτρια που έδωσε έμφαση σε δύο πτυχές που είναι ουσιώδες. Η διαφάνεια καταρχήν και η ε, de l'expertise, qui sont qualité et neutralité. Και ανεξαρτησία φυσικά. Αυτοί είναι δύο προϋποθέσεις ε, ε, απαραίτητες. Συμμερίζουμε φύσης ε, τη, όλες σφαιρικά τις απόψεις της ηγήτριας για το πρόγραμμα προετοιμασίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μέλη και θα πρέπει δηλαδή να δούμε ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει δικό της τρόπο ε, σύστημα αξιολόγησης τώρα θα πρέπει να είναι τέτοια τα συστήματα τα οποία θα πρέπει να είναι, όπου θα έχουμε διαφάνεια και να εξασφαλίζουν όλες τις προϋποθέσεις, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Θα πρέπει να δώσουμε μεγάλη έμφαση στο θέμα της ενεργασίας, να μπορούμε να προβλέπουμε τον κίνδυνο, να προλαμβάνουμε μια ε, πανδημία. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η έκθεση στο τέλος να δεχτεί την καλύτερη δυνατή, την πιο ευρεία υποστήριξη και να δοθεί έσφαση σε κάποιες πτυχές όπως η συν, ε, ο συντονισμός σε θέματα που φορούν την υγιεινή. Ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Κόνιντε Πάζα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε... πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για αυτή την έκθεση. Συμμερίζομαι πλήρως το, τις απόψεις της. Θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση. Καταρχήν, διότι μας επιτρέπει να έχουμε ανοιχτέ συζητήσει ειλικρινεί. Συμφωνείτε κύριε Πρόεδρε. Επίσης, μπορέσαμε να κάνουμε ερωτήσεις που δεν θα μπορούσαμε σε κάποιο άλλο διαφορετικό πλαίσιο να τις θέσουμε. Όπως τα θέματα που αφορούν τη διαχείριση και την ε, σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό ήταν το πρώτο σημείο. Δηλαδή ένα διαφορετικό τρόπο συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τι υπηρεσίε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μπορούμε να πάμε μακριά. Δεύτερο θέμα, όπω ελέγχθη από την Ντελμπού, ε, ότι είναι σημαντικό να λειτουργήσουμε καλύτερα συλλογικά και με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μα. Δεν γίνεται να προχωρούν οι χώρε μέλη ανεξάρτητα. Δεν είναι σωστό αυτό ε, δεν είναι σωστό ούτε για την αξιολόγηση ούτε για την παραγγελία εμβολίων διότι είναι χάσιμο πόρων. Ξέρουμε πόσο κόστισε αυτή η ιστορία στην Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό αποτελεί ένα μάθημα, για, μάθημα για όλους. Δηλαδή να προχωρήσουμε σε μια καλύτερη συλλογική ε, συνεργασία και προσέγγιση τόσο για την αξιολόγηση δεν, είναι, δεν έχει νόημα 27 διαφορετικές υπηρεσίε να κάνουν αξιολογήσει, αν είναι δυνατόν. Αυτό δεν εξυπηρετεί καθόλου. Και η τρίτη πτυχή είναι το θέμα που ετέθη για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι υπηρεσίε μας. Είναι ένα πιο ευρύ θέμα. Έχουμε να κάνουμε την οργάνωση όσον αφορά την εμπειρογνωμοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είδαμε κάποιε δυσκολίε με, την, ε, με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μολυσματικών Νόσων, Φερπίν. Το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Θεωρώ λοιπόν ότι θα ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτή η εντολή να προσθέσει, να δείξει, να επικεντρώσει το βάρος της σε συγκεκριμένους στόχους και θα δούμε το θέμα πώς λειτουργεί η εμπειρογνωμοσύνη. Είναι θεμελιώδος όσον αφορά την εμπιστοσύνη. Όλοι οι συνάδελφοι υπογραμμίζουν αυτό το θέμα. δεν είναι μόνο το θέμα των επιστημονών, των επιστημόνων. Ε, θα πρέπει παράλληλα να δούμε ούτω ώστε οι πολίτες μας από τη στιγμή που οι στην ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αξιόπιστοι ε, θα μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να προχωρήσουμε, να πάμε λίγο παραπέρα ε, όσον αφορά το γενικό συμφέρον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος. Τώρα Έχει έρθει ο ήδη και είναι έτοιμο να λάβει το λόγο. Ε, το αεροπλάνο μου, σας ζητώ συγγνώμη και επομένως δεν έχω παρακολουθήσει αυτά που είπαν οι προλαλήσαντες. Θέλω όμως να ευχαριστήσω την κυρία Ριβάση, η οποία επελήφθη με το θέμα αυτό της αξιολόγησης για τον ιό H1N1 είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια ισορροπημένη έκθεση για τα θέματα αυτά και σε αυτό μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι. Υπάρχουν πολλά ακόμα περισσότερα τα οποία θα πρέπει να διαλευκανθούν πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στην έκθεση της κυρίας Ριβαζή κατά την άποψή μου. Εγώ δεν θέλω να έχουμε μια έκθεση η οποία δίνει την εντύπωση ότι είμαστε κι εμείς λομπίστες για την ε, ε, φαρμακευτική βιομηχανία και υποστηρίζουμε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να προωθούν τα εμβόλια. Εμάς μας ενδιαφέρει να γνωρίζει ο πληθυσμός <clears throat> ποια είναι η πραγματική κατάσταση και να ξέρει ότι υπάρχει πολλές φορές απόλυτη ανάγκη για εμβολιασμό. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε την ισορροπία μεταξύ της αναγκαιότητος και του λογικού της αντιμετώπισης μιας πανδημίας. Επίσης, στη διάρκεια αυτής της ε, πανδημίας υπήρξε ιδιαίτερη έμφαση που δόθηκε σε θανατηφόρα περιστατικά. Είναι απλό. Θα ήταν πολύ απλό να δει κανεί όμως ότι η εξέλιξη αυτής της ε, ε, πανδημίας δεν είχε ε, υπερβολικά θανατηφόρα αποτελέσματα. Αυτό ήταν απλό και επομένως εγώ νομίζω ότι θα ήταν πολύ καλύτερα να μπορούσαμε να έχουμε την παρακολούθηση αυτής της πανδημίας. Τελικά για το γεγονός ότι δεν χρειάστηκαν όλα τα εμβόλια τα οποία ήταν διαθέσιμα, ότι ήταν, ε, υπήρξαν αρκετά εμβόλια και δεν υπήρξε έλλειψη, αυτό πρέπει να το καταχωρήσω στα θετικά στοιχεία της αντιμετώπισης Επίση, είναι απαραίτητο στο μέλλον να σκεφτούν τα κρατημέλη σε συνδυασμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία, με ποιο τρόπο μπορούμε να προλάβουμε μελλοντικέ πανδημίε, ποιε αρμοδιότητε θα πρέπει να αναλάβουν τα κρατημέλη και πώ θα πρέπει να γίνει η κατανομή των αρμοδιοτήτων ώστε να μπορούμε να είμαστε όλοι εξοπλισμένοι ενώπιον μια επερχόμενη πανδημία στο μέλλον και όχι το κάθε κράτο να κινείται από αυτού οι οποίοι έχουν συμφέροντα αλλά να μπορούμε όλοι μα να δρούμε από κοινού και να εκπροσωπεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση τα 27 κράτη-μέλη με τα 500 εκατομμύρια κατοίκων τους. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η Μαρίνα Γιανακουδάκη έχει το λόγο. Good morning, Chairman. Um, Καλημέρα σας κύριε Πρόεδρε. Πέρυσι νομίζω ότι βρεχιδερθήκαμε σε πολύ δύσκολη θέση αν θυμάμαι καλά. Είχαμε πανικοβληθεί, είχαμε δημιουργήσει αυτή την ανεπίση, την άτυπη επιτροπή, διακομματική, πάρα πολύ καλό αυτό, προσπαθούσαμε όλοι να βρούμε μία λύση. Το ενδιαφέρον όμως ήταν ότι είχαμε διαφορετικές ατζέντε, αν θέλετε. Δεν είχαμε μόνο την πανδημία. Ε, ανησυχούσαμε και για άλλους τομείς, όπως ε, η, η διαφάνεια. Υπήρχε μια αντιφαρμακευτική, αν θέλετε, διάθεση. Ε, και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το θυμόμαστε όλοι, ότι το βασικό πρόβλημα ήταν η πανδημία εν γέννη, όχι μόνο των χείρων, των πουλερικών, οποιαδήποτε πανδημία. Σε μια τέτοια κατάσταση ο πανικός είναι μεγάλος, η πίεση είναι ακόμα μεγαλύτερη, οι κυβερνήσεις ε, ε, αντιδρούν υπερβολικά ενίοτε και ο τύπος έπαιζε ένα πολύ κακό ρόλο θα έλεγα. Εγώ είχα, ε, θα υπερψηφίσω αυτή την έκθεση γιατί η Μισελ έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά γιατί θα πρέπει να δούμε τις διαδικασίες, θα πρέπει να δούμε τον ρόλο των υπηρεσιών, των φορέων, των οργανισμών ε, και όχι μονάχα ε, του, των του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μετά, ε, Μετάδοσης και Ελέγχου, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων. Δώσαμε μάχη για να δημιουργηθούν. Άρα θα πρέπει να έχουν πιο στενέ σχέσεις ε, και μεταξύ μα. Θα πρέπει να δούμε πώς αντιδρούν τα κράτη-μέλη. Τέλο πάντων, σε όλα αυτά όμω θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο βασικό μα στόχο είναι πώ θα αντιμετωπίσουμε ένα τέτοιο περιστατικό ξανά, αν παρουσιαστεί. Διότι θα ξαναπαρουσιαστεί και θα πρέπει να παραμερίσουμε τα θέματα που μας απασχολούν και να δούμε πόσο θα δράσουμε έγκαιρα, λογικά και συντονισμένα. Διότι τελικά δεν νομίζω ότι οι ιοί αυτοί γνωρίζουν σύνορα, άρα θα πρέπει να μπορέσουμε να δράσουμε διασυνοριακά, ενωμένα, σε όλη την Ευρώπη. Άρα θα ήθελα να υπερψηφίσουμε την έκθεση αυτή και θα ήθελα ε, όλοι να μην σκεφτόμαστε αυτά τα, τα δικά μας μόνο, αλλά να δράσουμε πιο ενωμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας χειροκρότησαν τα μέλη της ομάδας σας, πολύ καλό αυτό, να σας επικροτούν οι, συνεργά... οι συνάδελφοί σας. Η Άννα Ρόσπαχ δεν είναι παρούσα. Η Φρανσουάς Γκροστές λοιπόν έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε. Αυτό που θα ήθελα να σας πω είναι λίγο διαφορετικό από αυτά που ακούσαμε. Λυπάμαι που το λέω. Παρόλο που το έχω σεβασμό για τη συνάδελφο μου, όταν διαβάζω την έκθεσή της, δείχνει μία ε, έλλειψη ε, εμπιστοσύνης, πνευματική. πνευματικής. Ε, έχουμε τα θέματα ε, υγεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτήν την έκθεση βλέπουμε ότι ε, ενισχύεται το επίπεδο ε, έλλειψης κατανόησης και χωρίς να υπάρχει βάση. Σήμερα ξέρουμε ότι η πανδημία ήταν λιγότερο σοβαρή από ό,τι φοβόμασταν. Ε, και αυτό είναι πολύ καλό. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, αυτό να μην μας οδηγεί σε μια κατάσταση να σκεφτόμαστε ότι υπήρχε ε, και ότι ο, ΠΟΗ είχε κάποιες... δεν ήταν τόσο βέβαιος για τις επιπτώσεις. Είχαμε τη Γενική Διευθύντρια το 2009 είχε πει, ε, ε, έλεγε ότι ότι υπήρχαν κάποιε αμφιβολίε όσον αφορά τη σοβαρότητα αυτή τη ε, πανδημία, αλλά αυτό δεν είναι σωστό. Σίγουρα αποδείχτηκε ότι δεν ήταν τόσο σημαντική όσο φοβόμαστε. Η Ευρώπη προσπάθησε να προλάβει έναν κίνδυνο το οποίο δεν μπορούσε να εκτιμήσει εκείνη τη στιγμή. Αλλά αυτό που ισχύει είναι η αρχή της ε, πρόληψης. Και όλοι μιλάμε για αυτήν εδώ την αρχή και ξαφνικά σε αυτή την περίπτωση δεν έπρεπε να εφαρμοστεί. Ε, όλα αυτά τα εκατομμύρια που, που ξοδευτήκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη Γαλλία. Ε, αλλά είχαμε μια έκθεση λεπτομερή από το Υπουργείο ε, σε θέματα υγείας που δείχνουν ότι η εκτίμηση των εξοδεύτηκαν 547 εκατομμύρια ευρώ. Να μην λέμε ότι θέλουμε. Τώρα, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσματικών Ονόσων, θα ήθελα να πω ότι υπάρχει φήμη ότι είναι μία από τι καλύτερε υπηρεσίε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό με σοκάρει. Είχαμε ακροάσει και είχαμε κάνει ακροασει με αυτό το κέντρο. Αυτό που είναι κατανοητό είναι αν θέλει κανεί να, να είναι αξιόπιστο μπροστά στου πολίτε, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι δημορφηθήκαν 22 εκθέσει από αυτό το κέντρο. Όλες αυτές οι εκθέσεις είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα τους. Υπάρχει διαφάνεια. Θα ήθελα λοιπόν παρακαλώ να μην διαδίδουμε ό,τι να είναι. Είναι σημαντικό θέμα, έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία και να μιλάμε και να αναπτύσσουμε αυτή τη θεωρία περί παρακαλώ μην το κάνουμε. Δεν είναι, ε, θα έλεγα, έντιμο. Euh, Ευχαριστώ πολύ ο διευθυντής του ΟΜΕΑ είναι, θα είναι παρόν του Οργανισμού Φαρμάκων θα είναι παρόν στην Επιτροπή μας, οπότε θα μπορεί να εκφράσει και αυτό στην άποψή μας. Ο Σιλμαριό είναι ο πρώτος άνδρας, ο οποίος Πανιό είναι ο πρώτος άνδρας επιτέλους, ο οποίος λαμβάνει το λόγο για να υπάρχει μια ισορροπία σεξουαλικού χαρακτήρα. Θα πρέπει να θα προσπαθήσω να είμαι κάπως πιο αντικειμενικός. Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να τα βλέπουμε έτσι όλα μαύρα και άσπρα. Ε, και αυτό το λέω για σας κυρία Γκροστέτε. όντως υπήρξε ένα πραγματικό πρόβλημα και θα πρέπει εν ηρεμία να το εξετάσουμε και θα ήθελα να χαιρετήσω καταρχάς την ε, ποιότητα της έκθεσης της κυρίας Ριβαζή διότι δείχνει πάρα πολύ καλά ότι υπήρχαν και υπάρχουν κάποιες λύσεις σε αυτά τα προβλήματα τα οποία ζήσαμε όχι μόνο εμείς οι αιρετοί του ε, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά το σύνολο των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε αυτή την πανδημία που είχαμε εξαγγείλει, ότι είχαμε ακούσει ότι θα ήταν μια καταστροφή για την ανθρώπινη υγεία και στην Ευρώπη και σε όλο τον πλανήτη, αλλά που τελικά δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Άρα θα πρέπει να δοθούν κάποιες απαντήσεις και όσον αφορά την αρχή της προφύλαξη, που είναι μια πραγματικότητα και θα πρέπει να επανακτήσουμε την αξιοπιστία μας και την αξιοπιστία και να επαναρθώσουμε την αξιοπιστία αυτής της αρχής της προφύλαξης διότι ακριβώς αυτό είναι το θέμα σε σχέση με, την, με τους πολίτες μας ότι θα πρέπει να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας θα πρέπει να κερδίσουμε ξανά την εμπιστοσύνη των πολιτών διότι θα υπάρχουν και άλλοι που θα μας χτυπήσουν στο μέλλον επομένως τίποτα δεν θα είναι χειρότερο από, την, από το να βρεθούμε ενώπιον μιας διαδικασίες και ενός μηχανισμού όπου στο τέλος όλοι οι πολιτικοί άρχοντες θα χάσουν και αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις θα, χάσουν, ε, θα έχουν χάσει την αξιοπιστία τους. Επομένως θα πρέπει οι οργανισμοί αυτοί, οι υπεύθυνοι να είναι ανεξάρτητοι να είναι πιο ευέλικτη, να υπάρχει μια ε, δυνατότητα νέας διαμεσολάβησης όπως λέει η κυρία Ριβαζή στην έκθεση. Άρα θα πρέπει οι υπηρεσίες μας, οι οργανισμοί μας να μπορούν σε σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να έχουν μια μεγαλύτερη ανεξαρτησία και να ε, έχουν ε, πληροφορίες στη διάθεσή τους από εμπειρογνώμονες που να είναι πιο αξιόπιστες. Και αυτό πρέπει να επιζητούμε εμείς ε, σαν ε, βουλευτές. Θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες προτάσεις απέναντι σε αυτούς τους οργανισμούς. Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια απέναντι σε αυτούς τους οργανισμούς ε, είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να εξασφαλίσουμε τη διαφάνεια. Επίσης, σαν ερετή, αν θέλετε, μέσα από τη διαδικασία της καθολικής ψηφοφορίας, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την, το κοινωνικό συμφέρον θα πρέπει να μπορούμε να ελέγξουμε αυτές, αυτή, αυτή την ανεξαρτησία των υπευθύνων φορέων και οργανισμών. Δηλαδή να μπορούμε να πούμε να εδώ υπήρξε μια σύγκρουση, ε, μια σύγκρουση συμφερόντων. Συγγνώμη. Ε, επίσης, ανάλογα με, την, το τι θα δούμε, θα μπορούσαμε να ε, καθορίσουμε και την χρηματοδότηση. Θα μπορούσε να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε οι πολιτικές υγείας να εφαρμόζονται σωστά από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η κυρία Αντώνια. Α, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Ριβαζή για την έκθεσή της, διότι στην Ιταλία φανταζόμουν όταν, φανταζόμουν την έκθεσή της, θα την φανταζόμουν κάπως νεφελώδη, κάπως έτσι ανεκτική, ε, αλλά τελικά είναι πολύ καλή έκθεση και τη συγχαίρω. Για το πρόβλημα αυτής της γρήπη, της πανδημίας ε, ή τα έναν ή ένα και για την προηγούμενη πανδημία της γρήπη των πουλερικών δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχουν τρεις βασικές τάσει. Η πρώτη είναι ότι τα πάντα θα έπρεπε να είναι δημόσια. Ε, όμως ε, πολλά μείνανε κρυφά και ό,τι δημοσιοποιήθηκε φαίνεται ότι είναι αποτέλεσμα χειραγώγηση. Όλες οι περιπτώσει αποδείχθηκαν μάλλον οι επιπτώσει δεν αποδείχθηκαν. Δεν ξέρουμε καλά ακόμα ποιο είναι ο αριθμό των θυμάτων, ε, τα χρήματα, η, η, αποτελεσματικ... αποτελεσμα... αποτελεσματικότητα του εμβολιασμού. Εκεί δεν ξέρουμε. Τελείως αδιαφανή τα συμβόλαια, οι τιμές, οι διαφορές των τιμών ανάμεσα σε κράτη-μέλη. Επίσης επικρατεί πλήρης αδιαφάνεια για τον αριθμό των εμβολίων που χρησιμοποιήθηκαν, που παρέμειναν σε κανένα κράτο μέλο και μην δεν τα κάνει η κυβέρνηση για αυτά τα εμβόλια τα οποία δεν χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης δεν ξέρουμε ποια είναι η αποτελεσματικότητα του αριθμού των εμβολίων που χρησιμοποιήθηκαν. Ξέρουμε ότι αγοράστηκαν 90 εκατομμύρια εμβόλια από τη Γαλλία, 8 εκ των οποίων χρησιμοποιήθηκαν. Τι να κάνουμε τώρα, τα υπόλοιπα, τα 84, τι να τα κάνουμε. Τι έγιναν, το 82 εκατομμύρια ξέρω πόσα ήταν το εμβολίο που, έγιναν, που παρέμειναν. Άλλη τάση τώρα, η δεύτερη τάση. Αφορά την πανδημία. Και εδώ έχουμε δύο διαστάσεις πρόκειται για γρήπη και δεύτερον αφορά την διαφάνεια και τη χειραγώγηση. Και η τρίτη βασική τάση αφορά τα αμφιλεγόμενα επιχειρήματα. Δεν πρόκειται για μια έκθεση που, είναι, που τάσεται υπέρ ή κατά της του εμβολιασμού. Εδώ μιλάμε για την διαφάνεια την, και την ευθύνη. Αυτή, αυτά είναι τα θέματα της έκθεσης. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να λέει στους ευρωπαϊκούς οργανισμούς ότι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο μέλλον όταν μας βάζουν όλους σε, αυτό το, σε αυτή την παγίδα ε, να χρησιμοποιούνται χρήματα κοινοτικά, ευρωπαϊκά χρήματα, χωρίς να είμαστε σίγουροι ότι χρησιμοποιούνται σωστά και ότι υπάρχει μια ουσιαστική προστιθέμενη αξία. Επομένως, αυτά όλα τα επιχειρήματα ε, χρησιμοποιήθηκαν καθαρά για εμπορικούς λόγους. Ο Χόρς του έχει το λόγο. Ο δεύτερος άνδρας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ ήδη εκπλήτωμαι πόσο γρήγορα χάνουμε τη μνήμη μας. Εμείς είχαμε ζητήσει να λάβουμε πληροφορίες στην Επιτροπή μας όταν ξέσπασε αυτή η γρήπη και είχαμε ζητήσει να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την προστασία του πληθυσμού. Και τι λέμε, τώρα λέγαμε ότι όλα αυτά ήταν αποτέλεσμα όσο ήταν ευλακίες και εγώ δεν μπορώ να δεχτώ μια τέτοια αντιμετώπιση. Εγώ σαν πολιτικός δεν μπορώ να δεχτώ μια συλλήβδην επίκριση όλων των επιστημόνων και το να θεωρήσουμε ότι υπήρχαν ε, αλότρια κίνητρα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τα επιστημονικά Ινστιτούτα. Αυτό το βλέπω σαν να είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. υπήρξε αυτή η έκθεση και βλέπουμε να υπάρχει μια ε, υποψία χειραγώγησης. Φανταστείτε όμως να μην υπήρχαν καθόλου εμβόλια και να μην υπήρχε καθόλου αντιμετώπιση. Τι θα είχε συμβεί τότε. Λοιπόν, τι θα μας λέγανε. Θα μας λέγανε ότι δεν έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό. Θα υπήρχαν τεράστιες ουρές μπροστά από τα φαρμακεία και τα ιατρικά κέντρα ανθρώπων που θα θέλανε να εμβολιαστούν και δεν μπορούσαν και θα μας κατηγορήσαν ότι αδιαφόρησαμε για την τύχη τους. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο έχει αποδειχθεί ότι υπήρξε κάποια χειραγώγηση, ότι υπήρξαν κάποια παιχνίδια. Εάν κάποιο το πιστεύει αυτό, θα πρέπει να παρουσιάσει κάποια επιχειρήματα και κάποια στοιχεία προ την κατεύθυνση αυτή. Επιστημό... Επομένως, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει μια τέτοια καταδίκη χωρίς να υπάρχουν επιχειρήματα καθόλου και στοιχεία. Εγώ νομίζω ότι το βασικό στοιχείο εκκίνησης της έκθεσης είναι σωστό. Ότι πρέπει να υπάρξει και μια αντιμετώπιση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει μια κοινή πολιτική υγεία. Θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχει κάτι τέτοιο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα κράτη-μέλη θα συνεργάζονται και θα έχουν μια καλύτερη συνεργασία μαζί τους, μεταξύ τους. Υπήρξε παραδείγματος χάρη το παράδειγμα αυτό των εμβολίων, τα οποία μπορέσανε να χρησιμοποιηθούν θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί σε άλλα κράτη-μέλη εάν υπήρχε μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Βλέπω λοιπόν στον τομέα αυτό να υπάρξει αρκετό περιθώριο για να βελτιωθεί η συνεργασία μας. Εγώ δεν θέλω όμως να συνταχθώ με αυτούς οι οποίοι θέλουν με ένα ιδιαίτερα λαϊκιστικό τρόπο να αντιμετωπίσουν την ε, κατάσταση που δημιουργήθηκε λες και ήταν μονάχα αποτέλεσμα χειραγωγής και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Η Εστέντε Λάγκε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα πρέπει να, είμαστε λίγο πιο ε, επιβλακτικοί και λίγο να δείχνουμε κάποια διπλωματία όσο αναζητούμε αυτό το θέμα. Ο, θα πρέπει αυτή η έκθεση να είναι επικοδομητική. Φυσικά όμως υπάρχουν κάποιες αντιφάσεις σε αυτή την έκθεση όπου αναφέρεται Φέρυπιν ότι ήξερε κανείς ότι αυτή η ασθένεια ε, ήταν πολύ επικίνδυνη, αλλά ότι ε, αρχίζουμε να συζητάμε να κάνουμε κάποιες αναφορές στη Γενική Διευθύντρια του ΠΟΕ της κυρία Τσάν εκτιμής που έγινε το 2009. Θα πρέπει κατά με να δούμε ότι όλα δείχναν ότι μπορούσαμε να έχουμε μια πανδημία. Αυτά που είπε η κυρία Τσάν είπε ότι υπάρχει κίνδυνος. Τότε δεν ξέραμε ακριβώς. Αν δεν κάνει τα στοιχεία, ξέρουμε πολύ καλά ότι ένας ιός ε, μπορεί να μεταλλαχθεί και πρέπει να προετοιμαστούμε. Αυτό το στοιχείο λοιπόν δεν το βλέπουμε στην έκθεση. Είναι πολύ σημαντικό σε σχέση με την προσέγγιση που θα έχουμε και ποια θα είναι η στάση μας. Ένα δεύτερο στοιχείο τώρα. Αν θέλουμε να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι εν ώψη πανδημιών, θα πρέπει να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και συμφωνώ εδώ με την εισηγήτρια όσον αφορά τα εμβόλια, αυτό που θα πρέπει να γίνει θα πρέπει να γίνει έξυπνα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είχαμε διαφορετικούς τύπους εμβολίων ε, που λίγαν ή όχι αργότερα ή πιο νωρίς όσον αφορά τι διαφορε... χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ένα τρίτο στοιχείο, αν θέλουμε πραγματικά να έχουμε ε, επικοδιομητική προσέγγιση σε αυτό το θέμα, θα πρέπει τότε να σκεφτούμε ε, τους πολίτες σε ευρωπαϊκό πεδίο, επίπεδο. Πολίτες οποίους εκπροσωπούμε, οι οποίοι επιθυμούν να έχουν απαντήσεις σε ερωτήσεις και δεν καταλαβαίνουν πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Πιστεύω μια έκθεση του Κοινοβουλίου μας θα πρέπει να εκτιμήσει το ρόλο των διαφορών ε, ε, υπηρεσιών και θα ήθελα να πω ότι εγώ φοβάμαι ότι ε, προσπαθούν μερικοί να δημαγωγήσουν, ενδεχομένως να θίξουν κάποια θέματα καθαρά από πολιτική σκοπιά. Αυτά δεν αφορούν τον πολίτη. Δεν έχουν ε, ανάγκη δημαγωγίας ή να δούνε τις πολιτικές αντεπαραθέσεις. Αυτό που θέλουν είναι συγκεκριμένα πράγματα. Μια παρουσίαση, μια αξιολόγηση, η οποία επιτρέπει να μπορέσει κανείς να καταπολεμήσει μια αντίστοιχη κατάσταση. Θα πρέπει να θέλουν να ξέρουν γιατί Φερρυπίν σε κάτω χώρε, στην Ολλανδία παίρνουν κάποια αλφα μέτρα, ενώ στη Γερμανία είναι διαφορετικά. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δράσει με ε, ε, βασικό γνώμονα την ε, δημόσια ασφάλεια και μια εναρμονισμένη προσέγγιση. Θα πρέπει στο μέλλον να είμαστε έτοιμοι και καλύτερα προετοιμασμένοι. Δηλαδή να συντονίσουμε καλύτερα τις δράσεις μας. Ευχαριστώ. Σόνικ. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Ριβάζη για την έκθεση την οποία μας παρουσίασε. Νομίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ώστε οι πολίτες μας να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να είναι σε θέση να προβούν σε μια πραγματική αξιολόγηση κινδύνου. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλοι περιμένουν από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να μπορούν να αξιολογήσουν σωστά τους κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από μια ενδεχόμενη πανδημία. Πιστεύω ότι πρώτα απ' όλα αυτό θα πρέπει να είναι ένα εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία θα πρέπει να είναι υπεύθυνη για τα θέματα αυτά. Τίθενται από την έκθεση της κυρίας Ριβαζή μια σειρά από από ερωτήματα. Και είναι ερωτήματα που θέτουν και οι Ευρωπαίοι πολίτε και περιμένουν από εμά τι απαντήσει. Θα πρέπει να δούμε και το ρόλο των μέσων ενημέρωση που ίσω διόγκωσαν υπερβολικά την κατάσταση αυτή, κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφευχθεί στο μέλλον. Όλα αυτά τα ερωτήματα για μένα λοιπόν είναι εύλογα και θεμητά. Αυτό το οποίο θέλουμε να εξασφαλίσουμε είναι να μην δημιουργηθούν υπέρμετροι φόβοι από την πλευρά των πολιτών και να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες θα έχουν εμπιστοσύνη στα ευρωπαϊκά και τα εθνικά όργανα. Δεν αρκεί μονάχα να υπάρχουν μαζικές αλλά αγορές ε, εμβολίων ή να τίθενται κατά μέρος χρηματικοί πόροι για την αγορά φαρμάκων και εμβολίων. Εντάξει, είναι μια έκθεση στην οποία όλοι μας έχουμε τη δυνατότητα να καταθέσουμε τροπολογίες, αλλά συγχρόνως πιστεύω ότι θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση στα ερωτήματα τα οποία θέτουν οι πολίτες μας. Το πιο σημαντικό ερώτημα είναι, ναι, υπήρξε ή όχι κάποια χειραγώγηση. Εμείς θεωρούμε ότι στη χώρα μου, τουλάχιστον στην Πολωνία, υπήρξε από την πλευρά των μεγάλων φαρμακευτικών εταιριών κάποια χειραγώγηση γιατί καταφέρανε να τα να μεταφέρουν την ευθύνη για, τα, για, τις, για παρενέργειες στο κράτος και όχι στον εαυτό τους. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρος. Κρήτον Αρσένης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισαγήτρια, την κυρία Ριβαζή, για την έκθεσή της. Είναι πολύ σημαντικό και να αξιολογήσουμε καλύτερα τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, που μας κόσε πολλά χρήματα σε μια εποχή οικονομικής κρίσης στην Ευρώπη και να δούμε πώς μπορούμε να αποφύγουμε την επανάληψη αυτών των σφαλμάτων στο μέλλον. Δεν είναι ρόδινες οι προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άμεσο μέλλον και συγχρόνως η κλιματική αλλαγή σημαίνει και μεγαλύτερη επιβάρυνση της γεωργίας και της δασοκομείας αλλά και μεγαλύτερη πιθανότητα ανθρωπίνων ε, πανδημιών ή εμπασφυρτώσει ε, ασθενειών που θα επηρεάσουν τον πληθυσμό. Και φυσικά όλα αυτά έχουν και επιπτώσεις στις οικονομίες των χωρών μας. Θα συμφωνούσα λοιπόν με όλους τους συναδέρφους που όπως και η συγγήτρια ζητήσαν να έχουμε καλύτερη εμπειρογνωμοσύνη, καλύτερα και σαφέστερα κριτήρια για το πώς ακριβώς αξιολογούμε αν κάτι είναι πανδημία ή όχι, να υπάρχει μεγαλύτερο συντονισμός και καλύτερη χρήση οικονομιών κλίμακος και φυσικά δεν θα πρέπει να έχουμε και πανικό ο οποίο δημιουργείται χωρί λόγο στον πληθυσμό. Ωραία, αυτέ ήταν οι παρατηρήσει των μελών τη Επιτροπή. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από την Κομισιόν να αναλάβει ε, τη Σκητάλη, ο κύριος Ντερίς, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Κομισιόν, θα λάβει τώρα το λόγο να κάνει τα σχόλια από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Κομισιόν θα ήθελα να ευχαριστήσει και την Επιτροπή αλλά και την κυρία Ριβαζή για την έκθεσή της. Πιστεύουμε ότι με την περίοδο αυτή μετά την πανδημία θα πρέπει να αντλήσουμε τα διδάγματα από όλη αυτή την κρίση για την ε, ΙΤΑ 1 ή 1 και να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη κρίση η οποία θα μας πλήξει κάποια στιγμή. Γι' αυτό θα πρέπει να αξιολογήσουμε και να μελετήσουμε όλα τα αποτελέσματα και τα διδάγματα από την ε, κρίση αυτή. Υπάρχουν ε, Κυρία Ριβάζη, κάποιες μελέτες και κάποια συμπεράσματα των εμπειρογνωμόνων που προσπαθήσαμε να τα εξετάσουμε, να τα μελετήσουμε και κατά κράτη-μέλη έχουν κάνει κάποιες μελέτες που είναι διαθέσιμες. Υπάρχουν δηλαδή αρκετές πληροφορίες και αριθμητικά στοιχεία που νομίζω ότι μπορούμε να μελετήσουμε προσεκτικά. Τώρα, για κάποια σημαντικά στοιχεία τα οποία είδα στην έκθεση. Κάποια θέματα τα θίξαμε ήδη. Π.χ. ας πούμε, ο, με, μηχανισμός ε, για την ε, ε, συλλογή των στοιχείων που αφορούν την πανδημία εξετάστηκαν πολύ προσεκτικά και θα ζητηθούν και στο επόμενο Συμβούλιο το Δεκέμβριο. Αυτές οι πρωτοβουλίες μας θα μας βοηθήσουν να δημιουργήσουμε νέους μηχανισμούς και νέες υπηρεσίες. Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες που μας βοήθηκαν στα θέματα απειλών της δημόσιας υγείας. Η Κομισιόν θα υποβάλει στο Κοινοβούλιο το τέλος, στο τέλος του 2011 ε, μια νομοθετική πρωτοβουλία, ένα νομοθετικό κείμενο, το οποίο θα μας ε, βοηθήσει να χρησιμοποιήσουμε και τις ε, νομικές, τη νομική βάση να μας βοηθήσει να κάνουμε κάποια πρόοδο και θα υποφεληθούμε και από την ε, νομική βάση που μας προσφέρει η συνθήκη της Λισαβόνας. Διότι αυτό το οποίο μας, ε, επίσης μας ενδιαφέρει είναι να βελτιώσουμε και την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών. Ήθελα να πω ότι έχουμε ανεξάρτητα τεστ για την αποτελεσματικότητα και οι μελέτες αυτές γίνονται από κάποιες δημόσιες αρχές και από ερευνητές. Αναφέρθηκε ένα μεγάλο project το οποίο αποτελεί, ε, συντονίζεται από τον ΙΜΟ που είναι τη μελέτη από τη, της βιομηχανίας και τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητικά για τον εμβολιασμό της γρήπης. Αλλά θα έχουμε και άλλα επιστημονικά πορίσματα σύντομα. Επομένως η Επιτροπή αυτή θα ε, από επιστημονικά δεδομένα. Επίσης, πώς εγκρίνουμε τα εμβόλια και όλα αυτά τα φαρμακευτικά σκευάσματα που μας προσφέρουν οι φαρμακοβιομηχανίες. Όντως, σε όλες τις χώρες η βιομηχανία προσφέρει οι πληροφορίες, όμως η αξιολόγηση των πληροφοριών αυτών γίνεται από ανεξάρτητες επιτροπές. Και ελπίζω ότι με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθούν ε, και όλες αυτές οι συγκρούσεις συμφερόντων και δεν θα υπάρχουν αμφιλεγόμενες περιπτώσεις. Ελπίζουμε ότι θα, θα επενδύσουμε περισσότερο στην έρευνα και στα εμβόλια. Στο στάδιο αυτό η Κομισιό δεν θεωρεί σκόπιμη την διαδικασία αξιολόγησης των φαρμακευτικών σκευασμάτων που προτείνονται σε κρίσιμες περιόδους. Πιστεύουμε ότι το σύστημα το οποίο ισχύει και το οποίο ήδη το έχουμε προτείνει και το έχει εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Τώρα, όσον αφορά την τελευταία παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Κομισιό και η σχέση μεταξύ των δύο, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχει δικούς της μηχανισμούς για την, για την, για την αξιολόγηση που κάνει στα διάφορα σκευάσματα ή στοιχεία κτλ. Στις 25 Απριλίου του 2009 κάναμε την πρώτη αξιολόγηση όταν ξεκινούσε η πανδημία και προσπαθούσαμε να συγκεντρώσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία μας ερχόντουσαν από, ε, από όλα τα σημεία του πλανήτη για να γίνει μια σωστή αξιολόγηση και να μπορέσουμε να δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες στους όσους έπρεπε να λάβουν την, τις αποφάσεις. Το ερώτημα είναι ποιος θα συνοντήσει, ποιος μπορεί να συντονίσει μια παγκόσμια κρίση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, προφανώς. Τώρα, για τη σύγκρουση συμφερόντων. Και οι υπάλληλοι της, των, επιτροπών, της Επιτροπής. Εμείς πιστεύουμε ότι το προσωπικό της Κομισιό δεσμεύεται από το καταστατικό. Υπάρχει ένας κανονισμός. Και εκεί ε, εμφανίζονται σαφέστατα ε, τα προβλήματα των, ε, της σύγκρουσης των συμφερόντων. Λοιπόν, τις επόμενες μέρες θα έχουμε περισσότερη σαφήνεια νομίζω και περισσότερες πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ρης. Ο καθηγητής Άγκους Νίκολ από το ICDC, το οποίο αναφέρθηκε ήδη. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να περιοριστείτε μονάχα σε τέσσερα λεπτά για να μας δώσετε τη δική σας γνωμοδότηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι καθηγητής Νίκολ και είμαι ο υπεύθυνο συντονισμού στο ECDC από το 2007-2005 εντεύθεν. Μπορείτε να διαβάσετε την δήλωση οικονομικών συμφερόντων εμού του ιδίου και των συνεργατών μου στην ιστοσελίδα του φορέα μας, αλλά θα βαρεθείτε τα μάλα διαβάζοντας αυτά τα πράγματα. Εμείς χαιρετίζουμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η έκθεση η οποία εκπονείται από την Επιτροπή σας. Εμείς θέλουμε να υποστηρίξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι και το καθήκον μας, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι έχετε στα χέρια σας ακριβή στοιχεία. Και αυτή τη στιγμή, παρά το γεγονός ότι η έκθεση περιλαμβάνει θετικές παρατηρήσεις, είναι ανακριβή σε μία σειρά σημείων. Ο συνάδελφος μου ανέφερε μερικά από αυτά τα σημεία και ένα από αυτά αφορά την ανεξαρτησία του ECDC. Εμείς κάναμε οκτώ εκθέσεις αξιολόγησης κινδύνου κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Εκδόθηκαν ήδη από την αρχή της έκρηξης της πανδημίας και βελτιώθηκαν στην ε, πορεία του χρόνου ανεξάρτητα από την ΠΟΗ και με την βοήθεια των εμπειρογνωμόνων και δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο με αυτέ τι εκθέσει στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Επίση υπάρχει το θέμα του αποτελέσματο των ενδεχόμενων παρενεργειών των ε, εμβολιών. Των εμβολίων. Εμείς έχουμε χρηματοδοτήσει μία σειρά για, τη, για μελέτες σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Οι περισσότερε εκθέσει ήταν θετικέ, ήταν πραγματικά πάρα πολύ αποτελεσματικά αυτά τα εμβόλια. Αυτέ οι εκθέσει μα εστάλησαν το Μάρτιο πέρσι και δημοσιεύτηκαν τον Απρίλιο στην ιστοσελίδα μας. Δυστυχώς δεν ξέρουν οι ευρωβουλευτές τι υπάρχει στην ιστοσελίδα μας. Εμείς θέλουμε να βοηθήσουμε την κυρία Ριβάση, η οποία μονάχα έχει αναφερθεί σε ένα από τα έγγραφα του οργανισμού μας. Νομίζω ότι εάν εξέταζε και τα υπόλοιπα θα ήταν πολύ χρήσιμο. Αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε και εν ώψη του μέλλοντος είναι ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα τα οποία θα πρέπει να αντλήσουμε Σίγουρα τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη ευκαμψία και ευελιξία, αλλά πράγματι υπήρξε μεγαλύτερη ευκαμψία από ό,τι στα αρχικά σχέδια. Τα αρχικά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μερών δεν ήταν τα καλύτερα δυνατά. Η απάντηση όμως και η απόκριση τελικά ήταν πολύ καλή. η συνεργασία επίση και ο συντονισμό σε προευρωπαϊκό επίπεδο ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι αντανακλάται στην έκθεση αυτή. Η Επιτροπή Ασφάλεια και Υγεία συνεδρίασε μια μεγάλη, ε, ένα μεγάλο αριθμό φορών και τα κράτη-μέλη μπόρεσαν να συμβάλλουν πολύ περισσότερο από ό,τι αναμενόταν. Εμείς τώρα ε, ζητούμε από τα κράτη-μέλη να δούμε τι έχουν ε, σε τι έχουν ε, καταλήξει υπομορφή αξιολόγησης για την ε, επιδημία αυτή, υπήρχαν πολλαπλές εμπειρίες και πολλαπλές αντιμετωπίσεις. Δεν υπήρξε δηλαδή μια ενιαία αντιμετώπιση στα κράτη-μέλη. Επομένω, η ECDC θα ήθελα να σας βοηθήσει για την έκθεση αυτή, αλλά κυρίως θέλουμε να πληροφορήσουμε καλύτερα τους ευρωβουλευτές στο μέλλον σε σχέση με τα θέματα αυτά. Και επανερχόμενος σε αυτά που είπε ο διευθυντή μα και ο πρώην διευθυντή μα, νομίζουμε ότι τα καταφέραμε πολύ καλά. Απλώ θα πρέπει να υπάρχει μια σωστή αναλογικότητα, γιατί η τελευταία πανδημία ήταν χειρότερη τον δεύτερο χειρό χειμώνα και όχι τον πρώτο χειμώνα και δεν θέλουμε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Θα μπορούσε να έχει συμβεί και αυτό ήταν και ο λόγος για πολλές από τις αποφάσεις που ελήφθησαν το, την άνοιξη του 2009. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Καθηγητά Νίκολ. Φυσικά είναι δημόσιο σύστοση. Θα, θα εξετάσουμε πιο προσεκτικά τα όσα έχετε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα σας. Και τώρα η κυρία Παρβάνοβα θέλει να θέσει ένα ερώτημα νομίζω. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση η οποία, γιατί πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ποιο είναι το αντικείμενο των μελετών. Διότι άκουσα για μελέτες για την αποτελεσματικότητα των εμβολιασμών. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ ρωτώ κατά πόσον από ε, ε, τη σκοπιά, την επιστημονική και την σκοπιά της δημόσιας υγείας, κατά πόσον υπάρχει μία μελέτη που αποδεικνύει την διαφορά ανάμεσα στον αντίκτυπο της, του εμβολιασμού και τον αντίκτυπο της, ε, της ανοσίας του πληθυσμού. Έχει, μελετήσει κανείς ε, την προστιθέμενη αξία αυτού του εμβολιασμού σε σχέση με την ε, ανοσία, τη γενική ανοσία του πληθυσμού που ήδη υπάρχει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Ένα από τα πράγματα τα οποία ήταν ε, μη αναμενόμενα σε αυτή την πανδημία αλλά κάθε πανδημία ενδιαφέρει, είναι ότι υπήρχαν άτομα τα οποία ε, παρουσίαζαν ανοσία, π.χ. άτομα της ηλικίας μου. Από τις ανεξάρτητες μελέτες όμως που έγιναν είδαμε ότι υπήρχε προστιθέμενη αξία. Δηλαδή υπήρχε ένα 70% παραπάνω πιθανότητες να μην αρρωστήσεις εάν έκανες το εμβόλιο. Εάν δεν έκανες το εμβόλιο και αν δεν είσαι ανήκες στην ομάδα που είχε την ανοσία, ανοσία τότε αντιμετώπισες μεγαλύτερους κινδύνους και κυρίως οι νέοι και οι, τα νέα και τα υγιή άτομα. Το οποίο δεν το, το είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν το συναντάμε ευρέως στην κανονική γρήπη. Εντάξει, εδώ η απάντηση στην κυρία Παρβάνουα και δίνω ακόμα τρία λεπτά στην εισηγήτρια για να απαντήσει και να κάνει τα σχόλιά της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους παρεμβαίνοντας διότι ακούστηκαν πολλές παρατηρήσεις, θετικές και κριτικές όμως αλλά θα ήθελα να απαντήσω επί της ουσίας, εάν μου επιτρέπετε. Ναι, όντως, ε, κυρία Γκροστέτ, να, να ε, σεβόμαστε την αρχή της προφύλαξης, αλλά όταν υπάρχει ένας ιός τον οποίο δεν γνωρίζουμε καλά, και ε, καλό είναι να ε, δημιουργούμε ένα σχέδιο πρόληψης για το μέλλον. Όταν μιλάω για την ευελιξία και την καλύτερη αξιολόγηση των κινδύνων, θα πρέπει να, να δούμε ότι είτε πρόκειται για τις Ηνωμένε Πολιτείε, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ή σε διάφορα άλλα κράτη όπως ε, η Αργεντινή, το Νότιο Ημισφαίριο όπου είχαμε κρούσματα, τον Μάιο έγιναν αξιολογήσεις κινδύνων και σε σχέση με τον ε, ιό, κυρία Ντελόγκ, ξέραμε ότι ο, ο ιός δεν επρόκειτο να μεταλλαχθεί. Άρα είχαμε κάποιες απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Επομένως το ερώτημα το οποίο θέτω είναι γιατί να μην είχαμε μεγαλύτερη ευελιξία, γιατί σε σχέση με τα δεδομένα που είχαμε δεν επαναθεωρήσαμε τα σχέδιά μας. Δεν είμαστε εναντίον του αρχή, της αρχής ούτε εναντίον των σχεδίων ε, πρόληψης και αντιμετώπισης. Αλλά εάν δούμε όμως ότι ο ιός δεν είναι τόσο επιθετικός, εάν δούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού το οποίο δεν χρειάζεται να εμβολιαστεί, γιατί να μην αναθεωρήσουμε τα σχέδιά μας. Εδώ δεν είμαστε καλοί. Όσον αφορά τώρα σε αυτά τα, ε, αυτή κίνδυνη συνωμοσία. Δεν, υπή, δεν υπήρχαν τέτοια είδου σενάρια συνωμοσία. Όμως λέω ότι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας δεν υπήρχε διαφάνεια σε αυτή την επιτροπή ε, του, κα, την κατεπίγουσα. Ποια ήταν τα μέλη, δεν τα ξέραμε. Και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να επανεξετάσει τα κριτήρια για την πανδημία. Δεν μπορούμε να έχουμε έναν ορισμό ο οποίος να στηρίζεται μόνο στη γεωγραφική εξάπλωση και όχι στον αριθμό των θανάτων. Αυτό είναι απαράδεκτο. Οι εμπειρογνώμονες είναι σίγουροι όλοι και μα το λένε ότι δεν μπορεί να έχουμε μια επανάληψη όσο να γίνει το 2009. Επίσης, όσον αφορά την διαφάνεια, είχαμε τέσσερις γνωμοδοτήσεις του διαμεσολαβητή, ο οποίος ζητούσε να δημοσιοποιηθούν κείμενα και έγγραφα για κάποια φάρμακα. Όχι μόνο για την ΙΤΕΝΑΝΙΕΝΑ. Άρα δεν, υπάρχουν, δεν υπάρχει διαφάνεια. Για το εμβόλιο, η κυρία Γιακάμπα είχε πει, σα υπενθυμίζω, ότι κανένα εμβόλιο δεν εγκρίθηκε με τόσα λίγα επιστημονικά δεδομένα. Υπήρχαν δηλαδή δηλώσει κάποιων υπηρεσιών. Και αυτό το οποίο ήθελα να πω είναι ότι για το Ευρωπαϊκό Κέντρο είναι ότι προφανώ δεν αμφισβητώ την αρμοδιότητα και τι ευθύνε του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την μετάδοση και τον έλεγχο των ασθενειών. Όμω, αλλά όλα αυτά τα δεδομένα δεν αξιοποιήθηκαν. Δηλαδή, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν τα ξέραμε. Επίσης, ρώτησα την προηγούμενη φορά και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί αυτό το Ευρωπαϊκό Κέντρο τον Ιούνιο ή τον Μάιο του 2010 δεν μας είπε ότι δεν υπάρχει πλέον πανδημία στην Ευρώπη. Γιατί δεν το είπατε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση την πεφωτισμένη σας γνωμοδότηση να πει σταματάμε ε, διαδικασία της πανδημίας στην Ευρώπη διότι δεν υπάρχουν πλέον ε, περιστατικά. Ακολουθήσατε όσα είπε ο Πόη και ο Πόη σταμάτησε την πανδημία τον Ιούλιο. Εμείς θέλουμε να είστε ανεξάρτητοι, αποτελεσματικοί, να ενημερώνετε την, το Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να είναι όντω πεφωτισμένη η γνωμοδότησή σα. Ωραία, λέει ο Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η έκθεση αυτή ήταν πολύ σημαντική, γιατί σίγουρα θα πρέπει να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για το τι λειτουργήσε σωστά και το τι δεν λειτουργήσε σωστά στην αντιμετώπιση της ΙΤΑ 1 1, ώστε να είμαστε προετοιμασμένοι για τις επερχόμενες καταστάσεις. Και εγώ γνωρίζω ότι η Κομισιόν θα παρουσιάσει το Δεκέμβριο μια έκθεση προς το Συμβούλιο και σκέφτεται ακόμα και να προβεί σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Φυσικά εκεί θα πρέπει να κάνει και το δικό του έργο το Κοινοβούλιο για τη διαλεύκανση των όσων συνέβησαν και να έχει και κάποιες συστάσεις για το μέλλον. Ευχαριστώ λοιπόν τη Μισελ. Η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 1η Δεκεμβρίου στις 12 το μεσημέρι. Ψηφίζουμε στην Επιτροπή μας τον Ιανουάριο και αν θέλει ο Θεός θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια το Μάρτιο. Ευχαριστώ πολύ. Και ερχόμαστε στο επόμενο σημείο που είναι η, ερώτηση της κυρίας Σάτου Χάση για την ε, τοξική λάσπη στην ε, Ουγγαρία. Ε, ίσως ε, η κυρία Χάση θέλει να επανέλθει και να παρουσιάσει και πάλι το ερώτημά της. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω, λέει η κυρία Χάση την ερώτησή μου γιατί είναι σε γραπτή μορφή. Απλώς θέλω να ακούσω την απάντηση της Κομισιόν. Ωραία, θέτουμε λοιπόν το ερώτημα προς την Κομισιόν. Αν θέλετε να απαντήσετε τώρα το ερώτημα της κυρίας Χάση. Ποια είναι η θέση της Κομισιόν σχετικά. Κυρία Βένιγκ. Καλημέρα. Το όνομά μου είναι Μαριάννα Βένιγκε και είμαι υπεύθυνη της υπηρεσίας στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος ε, για τα θέματα βιομηχανικών εκπομπών. Καταρχάς, ε, θα ήθελα να εκφράσω τη συμπάθειά μας προς τις οικογένειες των ε, θυμάτων Περάσαμε μία φάση όπου εφαρμόστηκε ο πρώτος μηχανισμός πολιτικής προστασίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης και νομίζω ότι έκανε πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Καθήκον μας είναι τώρα να πάμε και να δούμε τι συνέβη πραγματικά και γιατί συνέβη. Και θα ήθελα να απαντήσω εδώ και στα ερωτήματα της κυρίας Χάτη. Κατά πόσον ε, διαπιστώσαμε βίαση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Σε αυτή τη στιγμή, αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να συλλέξουμε όλες τις πληροφορίες που μπορεί να μας δώσουν οι Ουγγρικές αρχές, πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να δούμε κατά πόσον ε, έχει παραβιαστεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να απαντήσουμε. Υπάρχουν κάποιες οδηγίες και να τις, να αναφέρουμε. Οι οδηγίες για την διαχείριση των εξοριγμένων αποβλήτων, ε, ένας κατάλογος, ευρωπαϊκός κατάλογος καταβλήτων, όπως επίσης και η οδηγία για την ε, περιβαλλοντική ευθύνη ε, προσπαθούμε να συλλέξουμε όλες αυτές τις πληροφορίες. Είχαμε επαφές με τις Ουγγρικές Αρχές και έχουμε στείλει και μια ε, επίσημη επιστολή 21 Οκτωβρίου και περιμένουμε την απάντησή τους. Επίσης έχουμε θέσει ερωτήσεις ε, σχετικά με την εφαρμογή όλων αυτών των οδηγιών και εδώ ε, φτάνουμε και στο δεύτερο ερώτημά σας για το κατά πόσο θεωρούμε ότι υπήρξε και κάποιο πρόβλημα σχετικά με τις επιθεωρήσεις. Ε, βασικά λέω το ίδιο πράγμα. Αυτή τη στιγμή εξετάζουμε ή περιμένουμε τις απαντήσεις των Ουγγρικών αρχών για να δούμε κατά πόσον οι απαιτήσει για τις επιθεωρήσεις και τους ελέγχους που προβλέπουν οι διάφορες οδηγίες έχουν γίνει σεβαστές ή υπήρξε πρόβλημα εφαρμογής. Ελπίζω ότι αυτές τις ε, ε, απαντήσεις θα τις πάρουμε μέσα στα πλαίσια της επιστολής που στείλαμε στις 22 Οκτωβρίου. Άρα περιμένουμε απάντηση από τι Ουγγλικές Αρχές. Τελεία. Άλλο ερώτημα. Κατά πόσον η Επιτροπή, ε, θα δημιουργήσει μια task force για να αξιολογήσει τα θέματα της ε, καταστροφής στην Ουγγαρία. Καταρχάς ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η παρούσα νομοθεσία, διότι υπάρχει σημαντική και λεπτομερής νομοθεσία και ένα κομμάτι αυτής της νομοθεσίας θα τεθεί πλήρως εφαρμογή το 2012 όταν μιλάμε για τα εξοριγμένα απόβλητα. Ε, η μια άλλη οδηγία ε, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο που μας δίνει την δυνατότητα να επιβάλλουμε πιο αυστηρές προδιαγραφές και απαιτήσει. Αυτές οι απαιτήσει εμφανίζονται στις διάφορες οδηγίες και θα πρέπει να εφαρμοστούν και με την ανάλυση των απαντήσεων που θα πάρουμε από τις Ουγγρικές Αρχές θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να ε, καλύψουμε τα κενά και να ε, διορθώσουμε την κατάσταση με, σε συνεργασία με την, Ουγγρική, την κυβέρνηση. Τώρα, για το πώς αντιμετωπίζουμε παρόμοιες, ε, παρόμοιους χώρους στην Ευρώπη. Υπάρχουν έξι χώρες που εξορίσουν βοξίτη στην Ευρώπη. Αυτές τις πληροφορίες που έχουμε όσον αφορά τις ποσότητες ε, του εξορισόμενου βοξίτη ε, είναι εδώ και, τις έχουμε εδώ και λίγο καιρό. Περιμένουμε νέες πληροφορίες ενημερωμένες. Έχουμε μια γενική κατανόηση ε, και πληροφόρηση και ενημέρωση για το τις δραστηριότητες εξόρυξης Και η βιομηχανία έχει κάποιες τεχνολογικές ε, δυνατότητες. Έχουμε επίσης 10 εγκαταστάσεις, 10 εργοστάσια αλουμίνας που χρησιμοποιούν, όχι είναι 10, συγγνώμη, 9 Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, Ιρλανδία, Ρουμανία και Ουγγαρία προφανώς ε, που χρησιμοποιούν ευοξίτη τα αυτά οι μήνες. Τώρα, όσον αφορά το νομικό πλαίσιο για τις ε, κοινοτικές επιθεωρήσεις ε, που αφορούν το σεβασμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας ε, και να είμαστε σίγουροι ότι οι περιβαλλοντικές αυτές επιθεωρήσεις γίνονται ανεξάρτητα και ομοιόμορφα. Η νομοθεσία για τις επιθεωρήσεις θα αναθεωρηθεί υπάρχουν συστάσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Η μία σύσταση είναι να ανανεωθεί απλώς η σύσταση που υπάρχει. Η άλλη δυνατότητα να υπάρχει μια οριζόντια οδηγία ή επίσης θα μπορούσαμε να εισάγουμε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για επιθεώρηση σε, τομιακές, σε τομιακά νομοθετικά κείμενα όπου θα έχουμε ένα συντονισμό των διαφόρων εναλλακτικών λύσεων και να υπάρξουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις επιθεώρησης. Ε, σας ανέφερα, σας την οδηγία για τις, για τις μηχανικές εκπομπές που εγκρίθηκε χθε στο Συμβούλιο. Εκεί υπάρχουν ε, υποχρεωτικές επιθεωρήσεις. Επίσης υπάρχει και η οδηγία ε, για την, για τα, που αφορά την, τα εξορισόμενα απόβλητα και εκεί προβλέπονται υποχρεώσεις επιθεώρησης και η Κομισιόν τόσο ή άλλως βρίσκεται σε η Κομισιόν για την, να ενδυναμώνουμε την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη επανεξετάζουμε τις εναλλακτικέ λύσεις που μας προτείνει το άρθρο 14 ε, θέλουμε να υπάρχει ένας εναρμονισμένος υποχρεωτικός μηχανισμός και εξετάζουμε κατά πόσον τα χρηματοδοτικά, οι χρηματοδοτικές απαιτήσεις και τα ανώτατα ποσά τα οποία ε, προβλέπονται είναι σωστά ή κατά πόσον πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση. Ε, αυτή τη στιγμή το μελετάμε το θέμα, δεν μπορώ να σας δώσω οριστική απάντηση. Συνειδητοποιούμε όμως το πρόβλημα και το εξετάζουμε. Όσον αφορά τώρα την αναθεώρηση του καταλόγου για τα επικίνδυνα απόβλητα. Καταρχάς θα πρέπει να ε, δούμε ότι ε, θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι οι αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνε για το κατά πόσον μια ουσία ή ένα προϊόν ε, αντιμετωπίζεται σαν επικίνδυνο, απόβλητο ή όχι. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκό Κατάλογο υπάρχουν δύο δυνατότητες για την ταξινόμηση και η σωστή, το σωστό θα πρέπει να γίνει από το κράτος Και αυτό εξαρτάται από την σύσταση του απόβλητου. Εάν ε, μιλάμε για παραπροϊόν ε, αλουμινίου και δεν έχει παρά μόνο βαρέα μέταλλα ε, και άλλες επικίνδυνες ουσίες, τότε μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν είναι επικίνδυνο. Αλλά από τη στιγμή που συμπεριλαμβάνει επικίνδυνες ουσίες που προέρχονται από τις φυσικές ή χημικές επεξεργασίες, τότε θα πρέπει να ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο και μέσω της άδεια που πήραμε από την εγκατάσταση ότι το προϊόν ε, δεν έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο. Αλλά βέβαια μπορεί να υπάρξει κάποια μόλυνση από βαρέα μέταλλα, άρα ζητήσαμε από τις Ουγγρικές Αρχές να μας πούν γιατί ταξινόμησαν τις ουσίες αυτές, τα προϊόντα αυτά σαν μη επικίνδυνα, σαν αυλαβή. Θα αξιολογήσουμε την απάντηση των κυρικών Αρχών και θα πρέπει μετά να πάρουμε μία απόφαση για το κατά πόσον η ταξινόμηση αυτή ήταν σωστή ή όχι. I think uh, I have addressed all the questions that were asked uh, Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω για σε περαιτέρω ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες σας σε σχέση με το ερώτημα της κυρίας Ρετ, της κυρίας ε, Χάση. Έχουμε πρόβλημα τώρα ότι είναι 11, ε, δεν μπορώ λοιπόν... Δεν μπορώ να δώσω το λόγο και στους 10 οι οποίοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ίσως οι Ούγγροι συνάδελφοι μπορούν να περιοριστούν σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ο κύριος Τσαμπατζή και η κυρία Χάση θα μπορούσαν να κάνουν ίσως μία παρατήρηση. Και είναι πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο και δεν έχουμε τη δυνατότητα μέσα στο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας να το συζητήσουμε. Ο Γιάννος Άντερ είναι ο πρώτος ο οποίος ζήτησε το λόγο. Παρακαλώ να είστε σύντομος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θέλω να υποστηρίξω την ε, παρατήρηση που κάνατε ότι πρέπει η Επιτροπή μας να ασχοληθεί με το θέμα αυτό σε ένα μεταγενέστερο χρονικό σημείο χωριστά για το θέμα αυτό. Όλοι οι συνάδελφοι από την Ουγγαρία έχουν δείξει ενδιαφέρον και οι άλλοι συνάδελφοι επίσης. Αυτό το ζήτημα επίσης είχε επιπτώσει και σε άλλες χώρες εκτός της ε, Ουγγαρίας και οι κοινοβουλευτικοί από άλλες χώρες έχουν δείξει και αυτοί ενδιαφέρον. Η κυρία Χάση έχει θέσει ένα σημαντικό ερώτημα. Θα πρέπει οι κανονισμοί και οι ρυθμίσεις για τα θέματα αυτά να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει προστασία και επίσης ότι θα διαλευκανθούν τα θέματα αστικής ευθύνης. Τα εργοστάσια παραγωγής αλουμίνας στην Ουγγαρία είχαν εγκριθεί, είχαν πάρει την έγκριση λειτουργίας το 2005-2006. Αυτό υπό την προηγούμενη κυβέρνηση. Η τωρινή κυβέρνηση δεν έχει να κρύψει τίποτα και δεν έχει την ευθύνη για αυτά τα οποία έλαβαν χώρα. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω τώρα. Για να μπορέσει να διαλευκανθεί το θέμα της ευθύνης και για να μην υπάρχουν περαιτέρω ζημίες στο μέλλον, η Ουγγρική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει για το σκοπό αυτό μια ειδική επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο του εργοστασίου αυτού αλουμίνες. Για να μπορέσει επίσης να γίνει σαφές το ποιος έχει την πραγματική ευθύνη αποφασίστηκε να σταματήσει η λειτουργία του εργοστασίου ώστε να μπορέσει κανείς να διακριβώσει ποιε ακριβώ ήταν οι ζημίε που προκλήθηκαν προηγουμένως προτού δοθεί η άδεια επαναλειτουργία του εργοστασίου. Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου, η κυρία Γκέοργεβα ανέφερε ότι η Ουγγρική κυβέρνηση έκανε ό,τι ήταν δυνατόν αυτή τη χρονική στιγμή, τη στιγμή της καταστροφής, για να αντιμετωπιστεί αυτή η καταστροφή. Διαβάσαμε επίσης το αρμόδιο έγγραφο ότι 700.000 ε, κιμικών μέτρων επικίνδυνων ουσιών απελευθερώθηκαν στο περιβάλλον. Υπάρχουν ακόμα 130 άτομα τα οποία είναι στα νοσοκομεία και 7 έχασαν τη ζωή τους. Νομίζω λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση ουσιών ως επικινδύνων θα πρέπει να υπάρξει πράγματι μια αλλαγή της ταξινόμησης αυτών των προϊόντων του εργοστασίου και εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται πιο έντονη ρύθμιση και πιο αυστηρή αντιμετώπιση. Επίσης όμως κάτι το οποίο γίνεται σαφές για μένα τουλάχιστον είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δώσει κάποια υποστήριξη μεν σε χρηματοοικονομικό επίπεδο, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει τα απαραίτητα μέσα. Θα πρέπει λοιπόν να το τροποποιήσουμε αυτό και θα πρέπει να έχουμε ένα ταμείο ή κάποιο άλλο τρόπο να υποστηρίξουμε οικονομικά τέτοιες φυσικές καταστροφές. Ο κύριος Ταμπάτζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έχουν δείξει αλληλεγγύη μαζί μας και μεγάλη προσοχή <clears throat> για, το, για τα προβλήματα τα οποία προήλθαν από τη φυσική καταστροφή που έπληξε την Ουγγαρία και είχε πολλά θύματα. Πρέπει να αντλήσουμε πολλά συμπεράσματα από αυτή την καταστροφή σε ό,τι αφορά την προστασία και του περιβάλλοντος. σε ό,τι αφορά την οδηγία <clears throat> περί ατυχημάτων. Νομίζω, περί βιομηχανικών ατυχημάτων. Θα πρέπει να γίνει πιο αυστηρή η αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. εξάλλου, υπάρχει και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες τόνοι ερυθράς λάσπης σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, στα, και στις χώρες των, των Βαλκανίων, στη Σερβία, Κροατία κτλ. Θα πρέπει να υπάρξει η απαραίτητη έρευνα για τις ε, ποσότητες αυτής της λάσπης που βρίσκονται στην Ευρώπη. Αυτό θα πρέπει να γίνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να αποτρέψουμε περαιτέρω καταστροφές. Εγώ συμφωνώ με την κυρία Χάση. Εδώ πρόκειται για την ανάγκη να έχουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή αντιμετώπιση και μια έρευνα η οποία θα πρέπει να γίνει σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να, κάνουμε μια, να δημιουργήσουμε μια επιτροπή η οποία θα διακριβώσει από πού προέρχονται οι ευθύνε για αυτό το γεγονό. Πέραν των Ούγγρων εμπειρογνωμόνων θα πρέπει να υπάρχουν και εμπειρογνώμονε από άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ούτω ή άλλω αυτό το οποίο είναι σαφέ, αυτό το οποίο έγινε σαφές ότι μια τέτοια, ένα τέτοιο ατύχημα θα έπρεπε να είχε αποφευχθεί και θα έπρεπε οι ουσίες οι οποίες προήλθαν από το ατύχημα να είχαν ήδη χαρακτηριστεί στο παρελθόν ως επικίνδυνες. Για το μέλλον επίσης θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να επαναχρησιμοποιήσουμε την ερυθρά λάσπη αυτή. Το θέμα αυτό δεν έχει επιληθεί ακόμα. Εγώ είχα θέσει ένα ερώτημα και η απάντηση της κυρίας Τζόρτζεβα ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα να επανα, επανα, ε, επεξεργαστούμε αυτή την ερυθρά λάσπη η οποία περιέχει ορισμένε επικίνδυνες ουσίες όπως είναι το τιτάνιο κτλ. Το πρόβλημα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης της ερυθράς λάσπης με τις τωρινές τεχνολογίες. Επίσης, τίθεται και το θέμα αυτό της χρήσης του Ταμείου για τις φυσικές καταστροφές που προς το παρόν δεν υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια για την αντιμετώπιση τέτοιων φυσικών καταστροφών. Έχουμε πάρει βοήθεια από όμορες χώρες όπως είναι η Σλοβακία αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο καλά λόγια και συμπαράσταση. Φυσικά πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και η εταιρεία η οποία προκάλεσε την φυσική καταστροφή. Θέλω ευχαριστήσω επίσης και την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ζήτησε να υπάρχουν να συμβάσεις ασφαλιστικού χαρακτήρα από τις εταιρείες αυτές τις εξορυκτικές και μεταλλουργικές και θα πρέπει να δούμε ποιο θα χρηματοδοτήσει εργασίε εκαθάριση. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι. Σα είπα ότι έχουμε αλλού οκτώ οι οποίοι θέλουν να λάβουν το λόγο, αλλά δεν υπάρχει καμία δυνατότητα να τους δώσω το λόγο. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησία διάταξη. Εξάλλου το θέμα αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσει ενδελεχέστερα η Επιτροπή μας. Θα επανέλθουμε λοιπόν εν καιρό και προς το παρόν περνάμε στο επόμενο σημείο της σημερινής διάταξής μας. Έχουμε την ε, πρέσβη ε, Σάνδρα Φουέντες από το Μεξικό μαζί με, τους εμπειρο... μαζί με τον... τους εμπειρογνώμονες της... για τα θέματα κλιματικής αλλαγής και είναι ενώπιόν μας γιατί όπως ξέρετε θα λάβει χώρα σε λίγες εβδομάδες η μεγάλη συνδιάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στο Κανκούν του Μεξικού. Το Μεξικό έχει προετοιμαστεί πολύ καλά. Θα γίνει και μια συνάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο κοινοβουλευτικών στο Μεξικό για τα θέματα αυτά και μετά θα ακολουθήσει η συνάντηση των εκπροσώπων των κυβερνήσεων που θα διαρκέσει δύο εβδομάδες. Γνωρίζουμε όλη τη Ελλάδα χώρα στην ε, Κοπενχάγη που δεν, δεν έδωσε θετικά αποτελέσματα για τα προβλήματα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και τώρα οι ελπίδες μας έχουν αναποτεθεί στην Μεξικανική Προεδρία και στη συνδιάσκεψη της Κανκούν από την οποία ελπίζουμε ότι δεν θα προέλθει πάλι αδράνεια και θα υπάρξει καν μια υποχώρηση σε σχέση με τις προηγούμενες δεσμεύσεις αλλά θα προκύψει πρόοδος και θετικά στοιχεία. Τα μέλη της Επιτροπής μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν ήδη αντιμετωπίσει ιδιαίτερα τα θέματα του περιβάλλοντος και έχουμε προετοιμάσει και ένα ψήφισμα βάσει του οποίου το οποίο θα πρέπει να εγκριθεί σε δύο εβδομάδες στο Στρασβούργο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήταν λοιπόν ενδιαφέρον να ακούσουμε από τη δική σας πλευρά ποια είναι τα κύρια σημεία στα οποία δίνει έμφαση η Μεξικανική Προεδρία Γνωρίζουμε ότι έχετε τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα θέματα αυτά, αλλά προφανώς και εσείς είσαστε πληροφορημένους για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρουσία σας στην Επιτροπή μας και θα ήθελα να σας δώσω το λόγο για να μας δώσετε τις ε, απόψεις σας και ένα, μια πρόγευση ουσιαστικά του τι αναμένεται από τη διάσκεψη της Κανκούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Γιολάινεν, Έχω μαζί μου ένα εμπειρογνώμονα για τα θέματα αυτά, γιατί φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν είμαι εμπειρογνώμο για τα θέματα, αλλά έχω ένα σύμβουλο από την Μεξικανική Πρεσβεία, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα αυτά και τον οποίο το γνωρίζετε και εσείς, γιατί ήδη έχει παρακολουθήσει και στο παρελθόν τα θέματα της κλιματικής αλλαγής από τη Μεξικανική πλευρά και εγώ επομένως θα λάβω το λόγο ενώπιον σας προφανώς, αλλά για ερωτήματα τα οποία θα απευθύνεται ιδίω αυτά που έχουν τεχνικό χαρακτήρα, θα τα παραπέμψω στον ε, σύμβουλό μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την ευκαιρία που μου δίνετε να λάβω το λόγο ενώπιόν σας, ώστε να μπορέσω να σας ε, παρουσιάσω ορισμένες από τις σκέψεις μας σε σχέση με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων για τα κλιματικά θέματα και σε σχέση με τα αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να προσδοκίσουμε από την διάσκεψη του Κανκούν, ώστε η διαδικασία της συμβάσεως πλαίσιου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή να μπορέσει να ανταποκριθεί στις πιο υψηλές προσδοκίες μας. Ξεκινώ αναφέροντας μια κάποια ανησυχία που ίσως ημερίζονται πολλοί από εσά. Οι πρόοδοι των διαπραγματεύσεων δεν ανταποκρίνονται στο επίπεδο γνώσης που έχουμε αυτή τη στιγμή σε σχέση με τις τωρινές και μελλοντικές προκλήσεις για την κλιματική αλλαγή. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι κατεπήγον να αντιμετωπίσουμε τα ενδεχόμενα αποτελέσματα αυτής της κλιματικής αλλαγής. Αυτό μας το λένε και οι μελέτες και οι προβλέψεις σε σχέση με το κόστος της αδράνειας στον τομέα αυτό. Υπάρχει μια γενική ανησυχία στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία των πολιτών, αυτούς οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα κινητοποιηθεί για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και οι οποίοι μας ζητούν να πάρουμε αποφάσεις που βρίσκονται στο ύψο των περιστάσεων και των προκλήσεων. Ούτε μπορούμε να επιτρέψουμε βέβαια στον εαυτό μας να απλοποιούμε τα πράγματα γιατί θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο πολύπλοκη είναι η, η πρόκληση και όχι να σταυρώσουμε τα χέρια. Πρόκειται για μια από τις πιο μεγάλες και τις πιο πολύπλοκες προκλήσεις που έχει αντιμετωπίσει ο Οργανισμός Εθνών λόγω της πολυπλοκότητας του θέματος και της αρνητικής πολιτικής και οικονομικής συγκυρίας αυτή τη στιγμή. Οι διαπραγματεύσεις αυτές λοιπόν ξεπερνάνε το απλό επίπεδο του περιβάλλοντος και ξεπερνάνε τις πραγματικές και σοβαρές ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή, γιατί περιλαμβάνονται και προκλήσεις που έχουν οικονομικό χαρακτήρα, ακόμα και προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ασφάλειά μας. Η μετάβαση σε μια οικονομία που καταναλώνει περισσότερο, που οδηγεί μάλλον σε μεγαλύτερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος δεν είναι μονάχα μια διεκδίκηση, είναι και μια πραγματικότητα και μια πηγή δημιουργίας νέων αγορών και θέσεων εργασία. που θα καθορίσουν σε μεγάλο βαθμό το επίπεδο ευμάρειας και ανάπτυξης όλων των χωρών στον κόσμο, ακόμα και θα επηρεάσουν και την ασφάλεια των χωρών αυτών στο μέλλον. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με την κλιματική αλλαγή σε όλες τις διαστάσεις της. Αν δεν ληφθούν οι απαραίτητες και ορθές αποφάσεις στην Κανκούν, κινδυνεύουμε αυτή την σημαντική διαδικασία να την κάνουμε μια διαδικασία που δεν θα έχει πραγματική σημασία για την κοινωνία μας και η οποία θα μπορέσει να χρονοτριβήσει για πολλά χρόνια, όπως δυστυχώς έχει συμβεί με τη διαδικασία της Ντόχα στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά μέσα σε ένα πολυετές πλαίσιο, ένα πολυμερές συγγνώμη πλαίσιο. Και το Μεξικό έχει δεσμευτεί να χρησιμοποιήσει όλη την ικανότητά μας και όλη μας τη διπλωματική μας εμπειρία για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία διαπραγματεύσεων και να έχουμε μια όσο το δυνατόν πιο φιλόδοξη απόλυξη στα θέματα της Σύμβασης για την κλιματική αλλαγή. Από το Tianjin βγήκε ένα κείμενο το οποίο θα ζητήσει μια ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια από τα κράτη-μέλη για να καταλήξουμε σε μια συνενετική λύση. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χάνουμε χρόνο σε παρελκυστικές διαδικαστικές τακτικές, ούτε να εμπλακούμε σε καθαρά ιδεολογικές ε, αντιμετωπίσεις και αντιπαραθέσεις βορανότου που έχουν δείξει τα όρια τους. Στην Κανκούν κάθε μία από τις εμπλεκόμενες πλευρές θα πρέπει να εντοπίσει τι είναι ουσιαστικό σε επίπεδο μεμονωμένο και να μπορέσει να προβεί σε παραχωρήσεις για το κοινό καλό να καταλήξουμε σε λύσεις που να είναι ικανοποιητικές γενικά. Το Μεξικό έχει κάνει ό,τι είναι δυνατό για να μπορέσει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη η οποία χάθηκε μετά από τη διάσκεψη της Κοπεχάγης. Έχουμε προχωρήσει σε μία σειρά από διαβουλεύσεις με όλες τις χώρες οι οποίες θα συμμετέχουν στην Κανκούν. Έχουμε κάνει προσπάθειες να συντονίσουμε τις ομάδες εργασίας και να χρησιμοποιήσουμε τις ε, υπηρεσίες διευκολυντών ώστε να καταλήξουμε σε ισορροπημένα αποτελέσματα. Όλο αυτό το χρόνο το Μεξικό προσπάθησε να προωθήσει και διάλογο μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών αρχών σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ε, χρηματοδότησης στην ε, Γενέβη τον αρχές Σεπτεμβρίου για την αγορά άνθρακος στη Βόνη τον Οκτώβριο και ένα τελευταίο επίσης ε, συνέδριο που αφορούσε τη χρήση τεχνολογιών. Και επίσης στην Κανκούν θα έχουμε και ένα χώρο εκθέσεων και διαλόγου όπου θα παρουσιαστούν πρωτοφουλίες ε, επιχειρήσεων, ε, προτάσεις για εμπόριο εκπομπών, προτάσεις για επενδύσεις στην αγορά του άνθρακα. Και εργαζόμαστε από στενά μαζί, συνεργαζόμαστε με το, Παγκόσμιο Συμβούλιο για τις εναλλακτικέ ε, ενέργειες και την κλιματική αλλαγή. Έχουμε λοιπόν προσπαθήσει να δημιουργήσουμε και κάποιο χώρο όπου θα συμμετέχουν οι ηθαγενείς πληθυσμοί. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάνω από 8.000 εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών που έχουν εγγραφεί στα Μητρώα βάσει των κειμένων ρυθμίσεων από τα Ηνωμένα Έθνη για να συμμετάσχουν στην COP16. Για τους φορείς τώρα που δεν θέλουν ή δεν μπορούν να καταγραφούν σε αυτά τα Μητρώα και να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του ΟΗΕ, η κυβέρνηση του Μεξικού δημιουργήσε και κάποιο χώρο όπου μπορούν να παρίστανται για να παρακολουθούν τις διαπραγματεύσεις. Είναι η λεγόμενη κλιματική πόλη, βίγια κλιμάτικα. Λόγω τώρα των συνθήκων αυτών και του λίγου χρόνου που έχουν στη διάθεσή μας, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Η πρώτη πρόκληση που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι αυτοί οι οποίοι θα παρίστανται στη Κανκούν είναι η έγκριση ενός πακέτου αποφάσεων που θα μας επιτρέψουν να διατηρήσουμε την διαδικασία διαπραγματεύσεων που θα οδηγήσει σε νομικά δεσμευτικές λύσεις και συμφωνίες τον επόμενο χρόνο. Θέλω εγώ να εκφράσω εδώ την ευγνωμοσύνη μου για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξει ένα δεύτερο χρονικό διάστημα για την επίτευξη δεσμεύσεων στα πλαίσια του πρωτοκόλλου του Κιώτο, που είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίω για τι αναπτυσσόμενε χώρε. Στην Κανκούν, είναι απαραίτητο να ενισχύσουμε το θεσμικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά τις προσαρμογές και τις ενσωμάτωσης τεχνολογιών που θα δώσουν μεγαλύτερη ικανότητα στις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Συγχρόνως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις αναγκαιότητες ε, βοήθειας προς τους πληθυσμούς αυτούς. Θα πρέπει να έχουμε ένα σωστό χρηματοπιστωτικό πλαίσιο το οποίο θα επιτρέψει να διοχετεύονται οι πόροι για τις αποτελεσματικές δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος τόσο σε ό,τι αφορά το μετριασμό των αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής όσο και μια μακροπρόθεσμη πολιτική αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε περαιτέρω ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίσει την διατήρηση των δασών και την αναδάσωση που έχει τόσο μεγάλα ωφέλη σε κοινωνικό και περιβαλλοντικό περιβάλλον. Θα πρέπει να προωθήσουμε και ένα σύστημα διεθνούς συνεργασίας το οποίο θα συμβάλλει στο να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί η ικανότητα σε όλες τις χώρες για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής και αυτό περιλαμβάνοντας και την μεταλαμβάνευση τεχνολογίας προς τους πιο ευάλωτους. Επίσης θα πρέπει να ενισχύσουμε και τις δράσεις μας μετριασμού των αποτελεσμάτων κλιματικής αλλαγής επί τη βάση των κοινών μας ευθυνών με τρόπο όμως διαφοροποιημένο επί τη βάση της ικανότητας κάθε χώρας τα θέματα τα οποία παρουσιάζουν μεγαλύτερε δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις είναι αυτά που έχουν να κάνουν με τις προσπάθειες μετριασμού τη κλιματική αλλαγή από τις αναπτυσσόμενες χώρες και τα θέματα που έχουν να κάνουν με την διαφάνεια η οποία θα πρέπει να αναφέρονται στην καταμέτρηση, την παρουσίαση εκθέσεων και την επαλήθευση των στοιχείων. Οι δράσεις μετριασμού από τις αναπτυσσόμενες χώρες και η απόδοση λογαριασμών έχουν ένα διαφορετικό νομικό χαρακτήρα από τις ε, ευθύνες και τις υποχρεώσεις που έχουν συνάψει οι αναπτυγμένες χώρες. Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε μια λύση, σε μια συμφωνία για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε σε σχέση με τις αποχρώσεις οι οποίες καθορίζουν τη διαφορά μεταξύ αναπτυσσομένων και αναπτυγμένων χωρών σε ό,τι αφορά την απόδοση εκθέσεων και λογαριασμών δεν πρέπει να σκεφτόμαστε για μεγαλεπίβολες αποφάσεις. Στην Κανκούν θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να καθορίσουμε ένα πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε στην, στο μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή που να οδηγήσει σε εθνικές δημόσιες πολιτικές που να είναι συμπεφωνημένες. Για να γίνει αυτό πραγματικότητα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια χρηματοδότηση η οποία μπορεί να δοθεί ταχαίως. Αυτό είναι θεμελιώδες αλλά επίσης θα πρέπει να πάρουμε και τι αποφάσει που θα επιτρέψουν τη δημιουργία του λεγόμενου πράσινου ταμείου που είχε συζητηθεί ήδη στην Κοπενχάγη. Η χρηματοδότηση δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι απλώ μία μορφή δώρων που δίνονται από τι αναπτυσσόμενες χώρε τι φτωχότερε, Είναι θέμα ισοδικία και δικαιοσύνη στον οικονομικό και περιβαλλοντικό τομέα επί τη βάση και της ιστορίας που έχουν γνωρίσει όλες οι χώρες μας. Επίσης είναι σημαντικό να μπορέσει να υπάρξει μια μείωση κατά 20 έως 30% των ε, εκπομπών αερίου θερμοκηπίου, όπως έχει αποφασίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 28 ε, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου 2010 αυτό θα γίνει μονάχα μετά από την Κανκούν. Η δική μου επιτροπή, η επιτροπή μάλλον της ε, της Κανκούν στο Μεξικό κάνει όλες τις προσπάθειες για να μπορέσει ο στόχο του 30% να προκριθεί έναντι του στόχου του 20%. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι είναι απαραίτητο να μειωθεί η θέρμανση της ατμόσφαιρας σε δύο βαθμούς μονάχα μέχρι το 2050. Αυτό στη συνέχεια θα πρέπει να τροποποιηθεί στο φως των νέων και εμπεριστατωμένων επιστημονικών στοιχείων. Αυτή τη στιγμή όμως δεν φτάνουν στο στόχο αυτό οι εθελοντικές ε, προσφορές για την μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου. Πρέπει λοιπόν όχι μόνο οι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι χώρε παρατήματο 1 και οι αναδυόμενες χώρες θα πρέπει να συμφωνήσουν σε πιο φιλόδοξους στόχους για τη μείωση της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου. Αυτό θεωρούμε ότι είναι εφικτό και το Μεξικό στρατηγικό εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξέρει ότι μπορεί να στηριχθεί στον ηγετικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ελπίζω θα μπορέσει να ασκήσει αυτόν τον ηγετικό ρόλο εναντί των εταίρων της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά εναντί και των χωρών οι οποίες λαμβάνουν βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθ' όλη τη διάρκεια λοιπόν αυτής της διαδικασίας είχαμε πολλές διαβουλεύσεις με σημαντικούς φορείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή ε, Επίτροπη φυσικά. Η Κόνη Χέντεργαρτ, η Επίτροπος Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στο Μεξικό και σήμερα ακόμα το πρωί μπόρεσα να ανταλλάξω απόψη μαζί της για τη σύνολη διαδικασία. Στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μιλήσει με μία μονάχα ενωμένη φωνή θα έχει μεγαλύτερο ειδικό βάρος. βάρος. Θα πρέπει να ασκήσει και μεγαλύτερη πολιτική επιρροή και πίεση σε χώρες με τις οποίες έχει σημαντικές ε, συνδέσεις εμπορικές και συνεργασίες. Το Μεξικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να λειτουργήσουν από κοινού. Να έχουμε τις απαραίτητες δομές συνεργασίας μέσα στα πλαίσια μιας συνολικής συμφωνίας. Έχουμε ήδη καταφέρει μέσα σε αυτό το κοινό να έχουμε 10 χρόνια καρποφόρων μορφών συνεργασίας. Θα πρέπει μέσα στα πλαίσια λοιπόν της COP16 ε, στη Κανκούν να συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία. Επίση όμω αυτό θα πρέπει να επεκταθεί και στι προσπάθειε για πιο καθαρή χρήση ενέργεια και πιο καθαρέ ενέργειε. Ελπίζουμε ότι οι προσπάθειε που έχουμε ξεκινήσει για μια παγκόσμια αγορά άνθρακο στο μέλλον θα μπορέσουν να οδηγηθούν σε σύγκληση με το σύστημα εμπορίας εκπομπών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι το πιο προχωρημένο στον κόσμο. Έχουμε ξεκινήσει ήδη διαβουλεύσει με την Κομισιόν για τη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθήσουμε και σε σχέση με τι κατατομής προοπτικέ Στο Μεξικό Είμαστε πεπισμένοι ότι πολλέ από τι λύσει οι οποίε θα πρέπει να δοθούν στα προβλήματα του περιβάλλοντο θα πρέπει να ξεκινήσουν από μηχανισμού αγορά. <clears throat> και γι' αυτό οι πολιτικέ μα προσανατολίζονται στο να δίνουν κίνητρα για μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην επίτευξη λύσεων. Ω χώρα που βρίσκεται στο παράτημα 1 του, του, του πρωτοκόλλου του Κιώτο, είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε περισσότερες δεσμεύσεις για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Όπως γνωρίζετε, ο Φελίπε Καλντερών στην αρχή του έτους έχει ανακοινώσει μονομερείς δεσμεύσεις για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου μέχρι το 2012 που είναι αντίστοιχες με 50 εκατομμύρια τόνων διοξιδίου του άνθρακος το χρόνο. Έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα δέσμευσης για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και έχουμε ήδη το θεσμικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία για να μπορέσουμε να αναλάβουμε ένα ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής και επίσης να είμαστε και τμήμα της νέας πράσινης οικονομίας του μέλλοντος. Το Μεξικό λοιπόν έχει φυσικά και την πλήρη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσει να προχωρήσει στην Κανκούν και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να προχωρήσουμε στην ουσιαστική ατζέντα και να ξεκινήσουμε μια νέα εποχή παγκοσμίων δράσεων για την κλιματική αλλαγή, για το καλό του Μεξικού, για το καλό της Ευρώπης και για το καλό όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Φουέντες για την παρουσίασή σας και για τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει το Μεξικό ως αμφιτρίωνας της ε, συνδιάσκεψης του ΟΗΕ και εγώ ίδιος ήμουν πριν από μερικές εβδομάδες στο Μεξικό και πραγματικά διαπίστωσα ότι υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον από όλη την κοινωνία του Μεξικού και μεγάλη διάθεση για συμμετοχή στην ε, διάσκεψη του, της Κανκούν και φυσικά η χώρα σας έχει αναλάβει ήδη μονομερείς δεσμεύσει ε, Είναι 8.000 ήδη οι εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών που θα θέλουν να είναι παρόντες και κατά πάσα πιθανότητα πολύ περισσότεροι. Ελπίζω ότι θα είναι καλή και η πρόσβαση στους χώρους της συνεδρίασης και όχι όπως στην Κοπενχάγη όπου έπρεπε κανείς να περιμένει πολλές φορές ώρες. Αναφερθήκατε επίσης και στις διαδικασίες διαπραγματεύσεων και την ανάγκη να τις ε, ε, βελτιώσετε. Είναι ουσιαστικά κατόρθωμα να μπορέσει κανείς να επιτύχει κάτι τέτοιο όταν υπάρχουν 193 ε, χώρες οι οποίες θα είναι παρόντες, παρούσες. Αυτό σε κάποιο βαθμό επετεύθηκε τότε στο Κιώτο πριν από δύο δεκαετίες και πρόσφατα πριν από δύο εβδομάδες στην Αγκόγια για τη βιοπικιλότητα. Όλα αυτά λοιπόν είναι δύσκολα αλλά εφικτά και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να απολύξουν σε αποφάσεις. Έχουμε μια μεγάλη σειρά λοιπόν από μιλητέ, Τρία λεπτά το μάξιμου σας παρακαλώ και δίνω καταρχήν το λόγο στον Καρλ Χάιτς Φρόρενς που είναι εδώ πέρα έξω δεξιά. Είμαι στην, ε, στην άκρη για να βλέπω τι πάει στραβά, ο κ. Καρλ Χάιτς Θέλω να καλωσορίσω την κυρία Πρέσβη και να την ευχαριστήσω με αυτά τα οποία είπε. Θέλω να σας ε, ενθαρρύνω να συνεχίσετε προς την κατεύθυνση αυτή της βελτίωσης της στρατηγικής μεταδιαπραγματεύσεων σε διπλωματικό επίπεδο και να λάβετε υπόψη ότι πολλές φορές είναι πολύ υπερήφανοι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων και εάν τους θίξει κανείς <clears throat> το κύρος τους κινδυνεύουν να πετάξουν από το παράθυρο όλα αυτά τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος. Πρέπει πιστεύω να λάβουμε υπόψη ότι ο δυτικός κόσμος πολλές φορές αντιμετωπίζει από αυτό το πρίσμα της ε, διαπραγματεύσης. Να απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάει με μια ενωμένη και ενιαία φωνή. Ο στόχος του, των δύο βαθμών μείωση της αύξηση θερμοκρασία είναι σημαντικό, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει πιο φιλόδοξα και να το μειώσει αυτό σε 1,5 βαθμό και μονάχα αύξηση τη θερμοκρασία μέχρι το 2050. Επίση, υπάρχει το περίφημο αυτό σύμπλεγμα του, της μέτρησης απόδοσης εκθέσεων και επαλήθευσης, το MRW. Αυτή η έννοια λοιπόν η οποία προέρχεται από την Κομπεχάγη. Πώς μπορεί κανείς όμως να τα πραγματοποιήσει όλα αυτά, δεν πρέπει αυτό να επιβληθεί με ένα αυταρχικό τρόπο σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό και πώς το βλέπουν και οι άλλοι εταίροι στα πλαίσια του ΟΗΕ. 1,5 βαθμός ε, μονάχα αύξηση θερμοκρασία, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο το εφήβρε η Επιτροπή μας, είναι όμως κάτι το οποίο ε, από την Κοπενχάγη, ήταν μια αίτηση πολλών χωρών, ιδίως νησιωτικών, οι οποίες με δύο βαθμούς αύξησης θερμοκρασίας κινδυνεύουν να μην υπάρχουν πια. Η Edith Εστρέλα έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω την κυρία Πρέσβη του Μεξικού και να την ευχαριστήσω για όλα αυτά που είπε και φυσικά να την ευχαριστήσω για τη δέσμευσή της ώστε η Κανκούν να είναι, αν δεν είναι επιτυχία, τουλάχιστον να μην είναι μια αποτυχία όπως ήταν η Κοπενχάγη. Αλλά συμμεριζούμε και εγώ τις δικές σας ανησυχίες. Γιατί αν είναι γεγονός ότι μετά από την αποτυχία της Κοπενχάγης έχουν μειωθεί οι προσδοκίες από την Κανκούν, εξακολουθεί να είναι γεγονός ότι οι επιστημονικές μελέτες μας κρούν τον κόνδυνα του κινδύνου και μας τονίζουν ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μεγαλύτερη πολιτική θέληση και μεγαλύτερη φιλοδοξία στον τομέα του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από την Κοπεχάγη, τουλάχιστον το Μεξικό φαίνεται ότι έχει αναλάβει τις ευθύνες του και το γεγονός ότι έχει δώσει και στην κοινωνία των πολιτών τη δυνατότητα να συμμετέχει, αυτό μου φαίνεται ότι είναι μια σωστή μεθοδολογία και ένας καλός ιονός. Είναι όμως απαραίτητο όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές να συμμερίζονται αυτό το αίσθημα ευθύνη και να υπάρξει καλύτερος συντονισμός και καλύτερη προετοιμασία για να μπορέσουμε να καταλήξουμε στα αποτελέσματα που όλοι ευχόμεθα να προκύψουν. Μας είπε πριν από λίγο ο πρόεδρος μας τα αποτελέσματα της συνδιάσκεψης της ε, Ναγκόγια για την βιοπικιλότητα. Όλα αυτά είναι καλά παραδείγματα τα οποία θα μπορούσαν να ακολουθηθούν και στην Κανκούν ώστε να μπορέσουμε να αποκομίσουμε θετικά αποτελέσματα. Αυτό το οποίο θα ήθελα επίσης να θέσω σε εσά ω ερώτημα μετά από αυτά που μας παρουσιάσατε είναι κάτι που έχει να κάνει με το λεγόμενο μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Ήμουνα πρόσφατα στο Εκουαδόρ μαζί με πολλούς άλλους ε, συναδέλφους από την συνέλευση Ευρωλάτ και είδαμε ότι υπάρχει μια κοινή θέληση χωρών της Λατινικής Αμερικής μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να δοθεί προτεραιότητα στα θέματα της, του μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. Θεωρείτε ότι είναι δυνατό να υπάρξει μια αρκετά φιλόδοξη συμφωνία για να δοθούν οι απαραίτητες επενδύσεις ώστε να μπορέσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες να προστατευτούν και να μετριάσουν την κλιματική αλλαγή. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η Σάτου Χάση έχει το λόγο. Όχι. Δεν θέλετε. Οι πράσινοι έχουν αλλάξει τους ομιλητές τους. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρέσβυρα για τις ε, πληροφορίες αλλά και για το ρόλο που παίζει το Μεξικό σαν ε, πρόεδρος αυτής της διάσκεψης. Και πιστεύω ότι και αυτό το που έκαναν οι Ιαπωνέζοι στην Αγκόγια θα σας βοηθήσει έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα και στο Κανκούν. Πρέπει να είμαστε σίγουροι όμως ότι ε, συνειδητοποιούμε ότι η τελική απόφαση δεν θα ληφθεί στο Κανκούν. Όμως θα πρέπει να γίνουν κάποια βήματα. Και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας και χαιρόμαστε που είσαστε διατεθειμένοι να κάνετε αυτά τα βήματα. Τώρα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το πώς βλέπετε εσείς την Ευρώπη να υλοποιεί το ρόλο της για το Κανκούν και κατά πόσον υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Διότι πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και αναφέρομαι πιο συγκεκριμένα στα θέματα για το εύρο του πρωτοκόλλου του Κιώτο για την πρώτη περίοδο. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αποκτά άλλο ένα και μεγαλύτερη σημασία για όλους Ποιο είναι το θέμα. Η Ευρώπη πάντοτε λέει ότι η περιβαλλοντική ακαιρεότητα του πρωτοκόλου του Κιώτο είναι ένα σημαντικό πρόβλημα και δεν μπορεί να διευρυνθεί. Όμως θέλω να ξέρω εάν εσείς θεωρείτε ότι η Ευρώπη είναι, θέμα, είναι κομμάτι του προβλήματος. γιατί η Ευρώπη αν θέλετε δημιουργεί, ε, ε, ε, δημιουργεί ναι, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Επομένως, εσείς κατά πόσον θεωρείτε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να παίξει έναν μεγαλύτερο ρόλο στην διατήρηση της περιβαλλοντικής ακεραιότητας του πρωτοκόλλου του Κιώτο και αν αυτό θα βοηθήσει περισσότερο το Κανκούνο; Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει και η κυρία Νταμπρά. Ε, θα ήθελα και εγώ να σας ευχαριστήσω, κυρία Πρέσβυρα, και για την δουλειά που κάνατε, γιατί έχετε, και το Μεξικό έχει μεγάλη διπλωματική ε, προϊστορία ε, και γνώση που θα χρησιμοποιήσει για να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο για το Κανκούν. Θα ήθελα να σας ζητήσω να μας δώσετε να, περισσότερες πληροφορίες για το πού θεωρείτε ότι βρίσκονται τα πράγματα και ποιες είναι οι σημαντικές αποφάσεις ε, για τη χρηματοδότηση και για το επίπεδο προσθετικότητας ε, όσον αφορά την χρηματοδότηση. Επίσης θέματα μεταφοράς τεχνολογίας ε, που υπάρχει το αδιέξοδο. Επίσης χαιρετίζω όσα είπατε για τα 8.000 ε, των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων που έχουν καταχωρηθεί. Ξέρετε ότι στην Κοπενχάγη πολλοί είχαν καταχωρηθεί, είχαν γραφτεί τέλος πάντων, αλλά όταν φτάσαν εκεί δεν μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τους υπευθύνους, δεν μπορούν να έρθουν ε, ε, σε επαφή με μας έτσι ώστε να υπάρχει αυτή η συζήτηση και η δημιουργία νέων, ειδών, νέων ιδεών. Επομένως θα υπάρχει δυνατότητα αυτής της φυσικής επαφής ανάμεσα σε όλους μας έτσι ώστε να ευδοκιμήσουν και οι ιδέες. Ο Ρίχαρτ Ζέμπερ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την ε, κυρία Φουέντες για τις ε, παρατηρήσεις σας. Το Μεξικό σαν ε, οικοδεσπότης έχει πολλές ευκαιρίες να μπορέσει να φέρει σε αίσιο πέρα σε αυτήν την ε, συνδιάσκεψη και να δείξει ότι τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν πράγματι να επιτύχουν πράγματι. Με ενδιαφέρε να ξέρω από την κυρία Πρέσβη τι ακριβώς προβλέπει να κάνει το Μεξικό υπό μορφή πρωτοβουλειών. Αναφερθήκατε ήδη το θέμα της ε, πράσινης οικονομίας και των ενεργειών και θα ήθελα να ξέρω αν το Μεξικό μπορεί να γίνει και αυτό μία από τις πρωτεύουσα της ε, δημιουργικότητος όπως η, η Βραζιλία έχει δείξει σε άλλους τομείς και η Νότιος Αφρική και επομένως να βοηθήσει τον αναπτυσσμένο χώρο την ε, Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες όπως και άλλες χώρες όπως η Κίνα που έχουν να διαδραματίσουν ένα ε, ιδιαίτερο ρόλο. Μετά από τις εκλογές ξέρουμε ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, η Κίνα δεν είναι ένας εύκολος εταίρος. Θα θέλω να ξέρω πώς θα μπορέσετε να πιέσετε τις χώρες αυτές να έχουμε περισσότερες κοινέ λύσεις. Ε, μιλήσατε για τη χρηματοδότηση και είπατε ότι το σημαντικότερο στοιχείο εδώ είναι η χρηματοδότηση startup για, την, για το ξεκίνημα των εγχειρημάτων και των συμπράξεων. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι τα συγκεκριμένα σχέδια τα οποία το Μεξικό προκρίνει για να, τυθού, να χρηματοδοτηθούν και ποιες είναι συγκεκριμένες για τι, ποιες είναι οι πρωτοβουλίες λοιπόν που εσείς θεωρείτε ότι είναι πιο σημαντικές και πώς θα πείσετε τους πολίτες ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει και χρηματοδότηση στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε την κυρία Πρέσβη για την παρουσίαση μας έκανε η οποία δίνει, θα λέγαμε, μας δημιουργεί μια αισιοδεξία. Ε, εγώ τώρα να σχολιάσω σε σχέση με τις δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να περάσει από το 20 μέχρι 30% μείωση μέχρι το 2020. Πριν από λίγο καιρό, σε μια πλειοψηφία είπαμε ότι θα μπορούσαμε να περάσουμε σε 30% στην Ευρωπαϊκή η Ένωση. Θα ξανασκεφτούμε πάνω σε αυτό το θέμα στην Ολομέλεια τον Νοέμβρη και θα εκφραστούμε σε ένα ψήφισμα για να δοθεί μια εντολή. Εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε από ακόμα περισσότερο. Ερωτήσεις. Όπως είπατε εξάλλου, υπάρχει πρόβλημα αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης κυρίως ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες και στις αναπτυγμένες χώρες, στις πλούσιες και τις φτωχές. Και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα το οποίο ήταν μεγάλο, όπως φάνηκε στην Κοπεχάγια. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι παραπάνω πάνω σε αυτό το θέμα, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ούτω ώστε να ξαναδημιουργηθεί ε, μια εμπιστοσύνη, ούτως ώστε να πετύχουμε μια συμφωνία ποιότητες. Και τώρα δεύτερη ερώτηση. Για τα στοιχεία που αναφέρετε, για τα συμπεράσματα που μπορεί κανείς να βγάλει από τη συνεδρίαση στο Μεξικό. Αναφέρετε τι θα ήταν απαραίτητο για να παρέχουμε επιτυχία ή αποτυχία. Ποια είναι τα κριτήρια επιτυχίας. Θα ήταν καλό ίσως να τα πούμε με σαφήνεια. Αυτά, α, β, γ, αυτά είναι τα κριτήρια που απαιτούνται. Η μη, άλλη μια φορά, θα μπορέσουμε να καταλήξουμε μια κατάσταση χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Εξάλλου έχει γίνει κάτι ανάλογο και στην Κοπεχάγη. Ευχαριστώ. Ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε και την κυρία Φουέντες για την παρουσία της. Θέλω να συγχαρώ το Μεξικό για το έργο το οποίο έχει φέρει σε πέρας μέχρι στιγμής. Αληθεύει το γεγονός ότι, ότι όπως είπε ο πρόεδρος μας ο κύριος Λάινεν, η επιτυχία σε δύο διοργανώσεις ήδη ανεβάζει τον πύχη αλλά θέτει και πίεση στις χώρες οι οποίες συμμετέχουν ώστε να υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα και φυσικά η χώρα που είναι οικοδεσπότης μπορεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο. Είναι γεγονός ότι αν δεν προχωρήσουμε, δεν πετύχουμε έστω κάποια πρόοδο στην Κανκούν, κάποια μικρή πρόοδο, μπορεί να καταλήξουμε σε ένα πλήρες αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν την Κανκούν μπορεί να καταρρεύσει το όλο σύστημα των διαπραγματεύσεων. Επομένω, είναι κομβικό αυτό το οποίο θα γίνει στο Μεξικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δούμε το αν θα μπορέσει μέσα στα πλαίσια του ΟΗΕ να υπάρξει μια συμφωνία για την κλιματική αλλαγή. Θέλω να σα θέσω το ερώτημα του αν θεωρείτε το αποτέλεσμα τη Ναγκόγια φέρνει ένα νέο ρεύμα στις, ε, στην πορεία των διαπραγματεύσεων, αν βοηθάει λοιπόν τα πράγματα. Και επίσης θέτω αυτό το ερώτημα, γιατί κάτι το οποίο διαπιστώσαμε στην Κομεχά είναι ότι όλοι πρέπει να κάθονται στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορούν να διαπραγματεύονται μόνο οι ισχυρέ χώρε και οι εκπρόσωποι των ομίλων χωρών. Όλε οι χώρε θα πρέπει να συμφωνήσουν, όλε οι χώρε θα πρέπει να βρίσκονται στι διαπραγματεύσει. Πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό στο Μεξικό. Πιστεύετε ότι χώρε όπω η Βενεζουέλα και η Μπολιβία δεν θα νιώθουν ότι έχουν αποκλειστεί από τις διαπραγματεύσεις και ότι θα συμμετέχουν πλήρως. Και ένα ερώτημα το οποίο έχει να κάνει περισσότερο με το μέλλον. Μήπως πιστεύετε ότι είναι πια καιρός να επανέλθουμε στο θέμα των χωρών του παρατήματος 1 και παρατήματος 2. Το 1998 όταν δημιουργήθηκαν αυτά τα παρατήματα η κατάσταση ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Τώρα έχει αλλάξει η συμβολή που μπορούν να κάνουν αυτές οι χώρες. Μήπως πρέπει στο Μεξικό, αν όχι αργότερα, να επανεξετάσουμε αυτό το θέμα και επίσης το Μεξικό θα είναι ενεργό και μετά την Κανκούν. Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό ο ρόλος σας τώρα, αλλά εμεί θέλουμε να διατηρήσετε αυτή την ενεργητικότητα και μετά την συνδιάσκεψη Κανκούν. Πάρα πολλές ερωτήσεις. Έχουμε άλλους δύο οι οποίοι θα λάβουν το λόγο. Ο Ζουάου Φερέρα έχει στη συνέχεια το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Πρέσβη για την παρουσίαση που μας έκανε εδώ και θέλω να θέσω εν συντομία δύο ερωτήματα εδώ. Σε ό,τι αφορά το μετριασμό, είπατε και πολύ σωστά πιστεύω ότι τα κονδύλια τα οποία θα πρέπει να δοθούν στις χώρες που είναι αναπτυσσόμενες για να υπάρξει ο μετριασμός και η προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές, ότι αυτά δεν είναι μια, ένα δώρο, ότι δεν είναι μια χορηγή απλώς, είναι ιστορική επανόρθωση για αυτά που έχουν κάνει οι αναπτυγμένες χώρες στο επίπεδο των αερίων θερμοκηπίων και την ανάγκη να αντιμετωπιστεί από όλους η χρηματοδότηση αυτή. Επίσης, τα ποσά τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση σχέδιων, το startup, το ταμείο αυτό της ταχείας εκκίνησης που αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όλα αυτά είναι πολύ λιγότερα από τα ποσά τα οποία θεώρησε απαραίτητα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι σε τάξη μεγέθους πολύ μικρότερα από αυτά που τα ποσά τα οποία συμποσούνται στο εξωτερικό, χωρών, στο εξωτερικό χρέος των χωρών αυτών. Είναι περίπου το ποσό αυτό περίπου μικρότερο από το 2% του εξωτερικού χρέους των χωρών της Ποσαχάριας Αφρικής το 2006 και το ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω εγώ είναι το εξής. Υπάρχει κατανόηση της ανάγκης να συνδεθεί το θέμα της χρηματοδότησης με την αντιμετώπιση του εξωτερικού χρέους των χωρών αυτών και είναι, υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει και η ακύρωση του εξωτερικού χρέους αυτών των χωρών λαμβάνοντας υπόψη την τεράστια πίεση που θα σημαίνει για τις χώρες αυτής οποιαδήποτε στρατηγική μετριασμού και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και στη συνέχεια αηφόρας ανάπτυξης. Το επόμενο ερώτημά μου έχει να κάνει με τους μηχανισμούς αγοράς. Λέτε κυρία Πρέσβη ότι θεωρείτε ότι οι λύσεις θα πρέπει να περάσουν και από την αγορά. Και αναφερθήκατε επίσης και στο ευρωπαϊκό σύστημα της εμπορίας εκπομπών που θεωρείτε ότι είναι το πιο προχωρημένο στον κόσμο. Κυρία Πρέσβη, στην πραγματικότητα το ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας εκπομπών, το οποίο ισχύει από το 2005, δεν οδήγησε στην πράξη σε μία μείωση της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου, κάθε άλλο οδήγησε στο αντίθετο αποτέλεσμα και είναι <clears throat> μία σαφής κατάδειξη του γεγονότος ότι οι μηχανισμοί της αγοράς δεν είναι αποτελεσματικοί. Το ερώτημα το οποίο θέλω να σας θέσω είναι κατά πόσο θεωρείτε ότι είναι απαραίτητο στην Κανκούν να τεθεί και το ερώτημα του αν μπορούμε να έχουμε μηχανισμούς εναλλακτικούς αυτών της αγοράς, λαμβάνοντας ακριβώς υπόψη τα όρια των μηχανισμών της αγοράς που είναι πρόδειλοι, όπως φάνηκε και στην περίπτωση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν είδαμε πόσο μετακινήθηκαν οι τιμές των εκπομπών άνθρακα μετά από την οικονομική κρίση. Μήπως λοιπόν στην Κανκούν θα πρέπει να συζητηθούν και άλλοι μηχανισμοί εναλλακτικοί με τους μηχανισμούς τη αγορά και να υπάρξει φυσικά και η συζήτηση για την αποτελεσματικότητα που είχαν μέχρι στιγμή οι μηχανισμοί της αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τέλος, η Σατουχάση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνεχίσω λίγο αυτά που είπε ο συνάδελφος. Ο, Αρκου, ο Ίσως ε, θα πρέπει να δούμε, να μας πείτε μάλλον εσείς, ποιες είναι οι απόψεις της μεξικανικής κυβέρνησης για το πώς θα μπορούσαμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στα θέματα χρηματοδότησης μετά τις κλιματολογικές διαπραγματεύσεις. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την καλύτερη δυνατή έκβασή τους. Πώς θα έχουμε μεγαλύτερη διαφάνεια στην ε, χρηματοδότηση έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ε, κλίμα εμπιστοσύνης στις διαπραγματεύσεις. Επίσης είναι γεγονός ότι δεν έχουμε μια συνολική συμφωνία εάν δεν θέλουν όλοι να αναλάβουν περισσότερες δεσμεύσεις. Αυτό ισχύει για τις βιομηχανικές χώρες, αλλά θα πρέπει και οι αναπτυσσόμενες χώρες να αλλάξουν τη στάση τους. Η μεξικανική κυβέρνηση τι κάνει για να δημιουργήσει ένα κλίμα θέλησης αν θέλετε από πλευράς των αναπτυσσόμενων χωρών ε, να αναλάβουν περισσότερη δράση, να αναλάβουν περισσότερες δεσμεύσεις στα θέματα κλιματικών αλλαγών να δεχτούν ας πούμε συνολικά όρια για τις εκπομπές ε, για το 2050 και ανώτατες, ανώτατα όρια εκπομπών. Ωραία. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις. Ήταν πολλές ερωτήσεις, οι οποίες έχουν θίξει μια μεγάλη, ένα μεγάλο φάσμα από ζητήματα. Βλέπω ότι σας έχει δώσει ορισμένα σημειώματα εμπειρογνώμων για να μπορέσετε να απαντήσετε. Είδατε ότι εδώ θέλουμε να είμαστε φιλόδοξοι από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή μας και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα έχει πιέσει την Κομισιόν και το Συμβούλιο να πράξουν περισσότερο γιατί έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι έχουμε μια μεγάλη ευθύνη έναντι του αναπτυσσόμενου κόσμου αλλά υπάρχει και το ερώτημα των ε, αναπτυγμένων χωρών και των χωρών κατοφλίου τι πρέπει να πράξουν. Από την εποχή του Κιώτο έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Η μετάβαση από το παράτημα 1 στο παράτημα 2, παραδείγματο χάρη, μπορεί να είναι ένα θέμα το οποίο κάνει ακόμα πιο πολύπλοκη τη στρατηγική διαπραγματεύσεων και επίσης τίθεται και το ερώτημα του τι βλέπει, ποια είναι τα κριτήρια που βλέπει το ίδιο το Μεξικό για την επιτυχία ή την απουσία επιτυχία στην Κανκούν. Και φυσικά και όλα τα άλλα τα ερωτήματα τα οποία σας έχουν απευθυνθεί είναι πάρα πολλά. Ελπίζω ότι μπορείτε να διεξέλθετε όλα αυτά τα ερωτήματα. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι πράγματι πολλές ερωτήσεις και πολύ ενδιαφέρουσες και ίσως δεν μπορέσω να τι απαντήσω όλες και σίγουρα όχι στη σωστή σειρά αλλά νομίζω ότι μπορώ να συμμεριστώ τις ανησυχίες όλων σας. Η... Όπως είπε και η Εντίτα Εστρέλα, υπάρχει και ένας κινησμός λιγάκι σε σχέση με την Κανκούν. Είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι δεν τρέφουν ιδιαίτερα υψηλές προσδοκίες μετά από την Κομπεχάγη που ήταν παρόντες όλοι οι αρχηγοί κρατών και είχε δημιουργηθεί ένα ιδιαίτερο κλίμα, μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα ότι ναι, επιτέλους θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα είναι νομικά δεσμευτική, η οποία θα επιλύσει όλα τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής κτλ. κτλ. Μετά από όλα αυτά, η Κανκούν δεν έχει ένα αντίστοιχο κλίμα και αντίστοιχες προσδοκίες. Ίσως είναι καλύτερα έτσι, γιατί αυτό το οποίο θα επιτευχθεί στην Κανκούν από μόνο του θα είναι πολύ πιο χρήσιμο για να προωθηθεί η διαδικασία αυτή διαπραγματεύσεων που όπως σας είπα προηγουμένως αυτή η διαπραγμάτευση πρέπει να γίνεται μέσα σε ένα πολυμερές πλαίσιο. Επίσης η ιδεολογική αυτή αντιπαράθεση βορανότου και ο αγώνας όπως αναφέρθηκε μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Όλα αυτά, όλοι αυτοί οι αγώνες δεν ξέρω αν βοηθούν σε κάτι. Όλοι ρηπαίνουν, ίσως όχι με την ίδια ποσότητα ρήπων και εκπομπών, αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε καταρχήν την ε, εμπιστοσύνη μεταξύ των ομάδων χωρών για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αναφέρθηκε το θέμα της διπλωματικής ικανότητας του Μεξικού. Το Μεξικό έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο μέσα σε πολυμερές πλαίσιο. Νομίζω ότι κατανοείται ότι λόγω της γεωγραφικής θέσης του Μεξικού η οποία γεωγραφική θέση δεν αλλάζει με τη διπλωματική δραστηριότητα, η θέση η γεωγραφική του Μεξικού μας υποχρέωσαν να έχουμε πάντα μια πολυμερή αντιμετώπιση ώστε να μπορέσουμε να υπερασπίσουμε τα συμφέροντά μας. Η εμπειρία λοιπόν του Μεξικού σε παγκόσμιο επίπεδο έχει σαν αποτέλεσμα να έχουμε επαφές και σημεία ε, σύγκλησης με πολλές χώρες του κόσμου. Είμαστε και εμείς οι ίδιοι σε μια ιδιαίτερη θέση γιατί είμαστε μια αναπτυσσόμενη χώρα αλλά είμαστε και μέλος του ΟΣΑ εδώ και 16 χρόνια, 15 χρόνια που θεωρείται η λέσχη των πλουσίων σε εισαγωγικά χωρών του κόσμου. Διατηρούμε λοιπόν ένα μόνιμο διάλογο τόσο με τον αναπτυσσόμενο κόσμο όσο και με τις αναπτυγμένες χώρες και νομίζω ότι μπορούμε να κατανοήσουμε τις ανησυχίες και των δύο ομάδων χωρών. Αυτό ήταν χρήσιμο και στην Αγκόγια όπου εμείς ήμασταν συντονιστές της ομάδας του Ρίο και από την άποψη αυτή νομίζω ότι έχουμε ήδη καταδείξει μέσα στη διάρκεια του 2010 το ότι έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε σε επαφή, να μιλάμε και να ακούμε όλους και να κατανοούμε τις ανησυχίες τους. Κάποιος έθεσε το ερώτημα του αν το Μεξικό μετά από την Κανκού θα συνεχίσει τις προσπάθειες αυτές. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Προεδρία μας ουσιαστικά ξεκινάει από την Κανκούν. Ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα το έχουμε κάνει σε ένα άτυπο, σε ένα ανεπίσημο επίπεδο. Πάντα με την υποστήριξη της Δανίας και την υποστήριξη της Νότιας Αφρικής δημιουργώντας έτσι με τη Δανία και την Νότια Αφρική ένα είδος τρόικας. Ελπίζουμε ότι φυσικά τα πράγματα θα προχωρήσουν και μετά από την Κανκούν. Από την άποψη αυτή μπορείτε να είστε σίγουροι ότι εμείς δεν έχουμε φυστεί προσπαθειών για να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, ότι θα είναι πλήρες και περιεκτικές αλλά κυρίω ότι θα είναι διαπραγματεύσεις που θα λάβουν χώρα σε ένα κλίμα διαφάνειας. Και εδώ θέλουμε να δώσουμε ένα παράδειγμα. Πιστεύω ότι ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων που έχουμε ήδη ξεκινήσει υπάρχει τουλάχιστον κάποια πρόοδο στη μεθοδολογία. Κάτι το οποίο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. λοιπόν αυτές που έχουμε καταβάλει θεωρούμε ότι θα μας οδηγήσουν σε θετικότερα αποτελέσματα στο μέλλον, ώστε οι χώρες οι οποίες θα αναλάβουν τη σκητάλη, θα αναλάβουν την Προεδρία, να μπορούν ήδη να ξεκινούν μετά από την προηγούμενη ε, συνδιάσκεψη. Θα μπορούσε παραδείγματο χάρη το Μεξικό να έχει αναλάβει την Προεδρία αμέσως μετά από την Κομπεχάγη και όχι το επόμενο έτος. Αλλά αυτό δεν είναι θέμα ουσία, είναι θέμα διαδικασία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε, θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα ισορροπημένο πακέτο σε όλα αυτά τα ζητήματα στα οποία υπάρχει ήδη μια συμφωνία και για τα οποία εμείς έχουμε συζητήσει εδώ και αρκετό καιρό με όλες τις χώρες και τις ομάδες χωρών. Σε ό,τι αφορά τις αναπτυσσόμενες χώρες, η στρατηγική μας ήταν να προσπαθήσουμε έτσι κάνουμε, να κατανοήσουν ότι η απάντηση στην κλιματική αλλαγή είναι από την ίδια τη φύση αλληλένδετη με τις πολιτικές ανάπτυξης. Επομένως πρόκειται για μια ενεξελίξη διαδικασία. Είναι φυσικά πολύ σημαντικές οι προκλήσεις, αλλά υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες οι οποίες ανοίγονται με την ε, διάσκεψη της Κανκούν. Κάποιος αναφέρθηκε σε κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα ε, για τη βοήθεια που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Μεξικό σε διαδικασίες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής εν Και μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ήδη ε, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ιδιαίτερα για πράσινα σχέδια, τα οποία έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούνται σε επίπεδο 50 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία χρησιμοποιούνται, 20 από τα οποία χρησιμοποιούνται καταρχήν για να χρηματοδοτηθούν σχέδια αιωλικής ενέργειας στη, στο κράτος της Οαχάκα, στο νότιο μέρος του Μεξικού. Είναι μια επαρχία που είναι γνωστή ως η ε, η επαρχία των αέριδων. <clears throat> Όλα αυτά λοιπόν είναι μια ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιχειρήσεις της να συμμετάσχουν σε επενδυτικά σχέδια αυτού του είδους και τονίζω επίσης ότι για μας ο διάλογος με τον ιδιωτικό τομέα παίζει ένα κεφαλαιόδη ρόλο. Εγώ ήμουν στο Μεξικό μέχρι πριν από δύο εβδομάδες, συναντήθηκα με ομάδες επιχειρηματιών και όλα αυτά τα οποία έλεγαν για τις κυβερνητικές πολιτικές ήταν ιδιαίτερα οδυνηρά. Θεωρούν ότι το κράτος τους κόβει τα φτερά, δεν τους επιτρέπει να αναπτύξουν επιχειρηματικές σχέσεις, ότι είναι απαραίτητο να κάνουμε πολλά περισσότερα, να συνεργαστούμε με τους γείτονέ μας, γιατί να περιορισμούμε λοιπόν τις δυνατότητές μας. Βλέπω λοιπόν ότι πάντα είναι απαραίτητο να κατανοήσετε ότι η κυβέρνηση του Μεξικού κρατάει μια υπεύθυνη στάση. Θεωρούμε ότι στο βαθμό που οι ιδιωτικές εταιρείες και ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να εμπλακεί με τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, θα έχουμε πολύ περισσότερες δυνατότητες να προχωρήσουμε. Οι πρόσφατες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις τεχνολογίες καθαρής και ανανεώσιμης ενέργειας θα μπορέσουν να βελτιώσουν την πρόσβαση σε σημαντικές πηγές χρηματοδότησης, οι οποίες σε τελική ανάλυση θα οδηγήσουν σε καθαρότερη και καλύτερη στέγαση, καλύτερες μεταφορές για τους πολίτες μας, σε λιγότερη εκπομπή ρήπων, σε λιγότερα αναπνευστικά νοσήματα, σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όλους και θα οδηγήσουν σε πιο αηφόρα χρησιμοποίηση της γης, των δασών, του ύδατος, όλων των φυσικών πόρων. Νομίζω λοιπόν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να εξασφαλίσουμε ότι η κλιματική αλλαγή θα είναι ένα εγχείρημα κερδοφόρο για τις χώρες του κόσμου. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος, Πιστεύω ότι το πολιτικό σκέλος θα πρέπει να συμβαδίζει με τις ε, ενέργειες ανάπτυξης και με τον τρόπο με τον οποίο η κάθε χώρα διαχειρίζεται τα εσωτερικά της οικονομικά θέματα για μένα. Ο τρόπος με τον οποίο θα ακολουθηθεί αυτή η πολιτική θα πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο σοβαρό και υπεύθυνο γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε ένα θετικό παράδειγμα και αυτά τα οποία είπε η κυρία Χάση είναι σημαντικά. Ρώτησε πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει, πώς είναι δυνατόν να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τις υπόλοιπε χώρες του κόσμου. Η απάντησή μου στο σημείο αυτό θα ήταν ότι πρέπει να διαδραματίσετε Ήδη έχετε ένα ηγετικό ρόλο. Δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ο ηγετικό σα ρόλο, αλλά τον έχετε. Πρέπει να συνεχίσετε να ασκείτε αυτόν τον ηγετικό ρόλο μέσα στα πλαίσια του, του, της Προεδρίας του Μεξικού. Εμείς συνεργαζόμαστε στενά με τις ευρωπαϊκές αρχές. Εγώ θεωρώ ότι η δική μας αγορά για τις εκπομπές ε, άνθρακα είναι ουσιαστικά ένα αντίγραφο του ευρωπαϊκού Συστήματο, Κάποιοι από εσά μπορεί να μην συμφωνείτε, αλλά αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι και ένα τρόπο με τον οποίο μπορούμε να καταλήξουμε σε ευρύτερα πρότυπα και σε πολιτικές οι οποίες θα αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Όλα αυτά είναι παραδείγματα τα οποία έχουμε πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Και προφανώ και το θέμα τη χρηματοδότηση θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο στι επόμενε ε, προσπαθίε μα. Δεν θέλω τώρα να εμπλακώ ιδιαίτερα σε τεχνικά θέματα, αλλά δεν χωρεί αμφιβολία ότι οι χώρε οι αναπτυσσόμενες χώρες περιμένουν χρηματοδότηση από τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου. Τώρα το ερώτημα του αν θα πρέπει να φτάσουμε στην ακύρωση του χρέους των πιο φτωχών χωρών. Και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο... Και αυτό θα πρέπει να συνδέεται με την ε, αποδοχή της ιστορικής ευθύνης που έχουν οι αναπτυγμένες χώρες για την κλιματική αλλαγή. Δεν πρέπει όμως να συγχαίουμε τα ποσά αυτά τα κονδύλια που δίνουν οι αναπτυσσόμενες χώρες για την κλιματική αλλαγή ως τμήματα μιας γενικής αναπτυξιακής βοήθειας. Είναι χωριστό θέμα η αναπτυξιακή βοήθεια και είναι χωριστά τα κονδύλια τα οποία είναι μια χρηματοοικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και για τις επιχειρήσεις ταχείας εκκίνησης. Υπάρχουν πολλοί στη διεθνή κοινότητα που λένε ότι αυτό πρέπει να το μετωπιστεί ως τμήμα της αναπτυξιακής βοήθειας. Εμείς όμως από τη δική μας οπτική γωνία δεν δεχόμαστε μια τέτοια αντιμετώπιση. Για τις ε, ΜΚΟ. Είναι πολύ σημαντικό να τονίσω ότι το Μεξικό θεωρεί πάρα πολύ σημαντικού εταίρους της ΜΚΟ στο διάλογο της Κανκούν. Θέλω όμως να σας υπενθυμίσω ότι οι κανόνες και η διαδικασία της ε, συνδιάσκεψης Κανκούν δεν καθορίζονται από τη μεξικανική κυβέρνηση. Εμεί είμαστε οικοδεσπότες. Εμεί δίνουμε το σπίτι μα για να οργανωθεί το πάρτι, αλλά το πάρτι δεν το οργανώνουμε εμεί, το οργανώνει ο ΟΗΕ. Επομένως η πρόσβαση στο ΜΚΟ θα πρέπει να ακολουθήσει το υπόδειγμα το οποίο έχουν καθορίσει τα Ηνωμένα Έθνη. Ε, αυτό το οποίο μπορούμε να του προσφέρουμε είναι καλύτερο καιρό από ό,τι στην Κοπενχάγη και ελπίζουμε και ο χρόνος αναμονής θα είναι μικρότερος, πάση δεν θα είναι στους μείον 20, αλλά μάλλον στους συν 30 που θα περιμένουν όσοι χρειάζεται να περιμένουν και φυσικά οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις θα έχουν πρόσβαση όχι στους χώρους όπου θα λαμβάνονται οι αποφάσεις, αλλά σε κάποιες αίθουσες όπου θα μπορούν να παρακολουθούν τα τεκτενόμενα. Φυσικά κάποιοι χώροι δεν θα είναι ανοιχτοί για τις για τις ε, ΜΚΟ όπως ε, πάντα γίνεται στα πλαίσια των συνδιασκέψεων του ΟΗΕ. Επίσης θέλω να εξάρω τη συμμετοχή των ηθαγενών πληθυσμών σε αυτή τη διαπραγμάτευση γιατί και αυτοί διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ελπίσουμε λοιπόν στην Κανκούν ότι θα είναι παρόντες 16.000 αντιπρόσωποι συνολικά. 16.000 μάλλον παρισταμένων. Εγώ μίλησα για 8.000 καταγεγραμμένες ΜΚΟ. Εσείς άμα κάτσετε και το υπολογίστε, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό συμμετεχόντων και καταβάλουμε μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να μην διαψευστούν οι προσδοκίες όλων αυτών όπως έγινε στην Κοπεχάγη όπου δεν είχαν ουσιαστικά καμία πρόσβαση στα τεκτενόμενα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει περίπου όλα τα θέματα τα οποία τέθηκαν. Θα ήθελα να σταθώ επίσης και στο θέμα της διαφάνειας που ανέφερε σαν του χάσει. Και αυτό είναι σημαντικό και θεμελιώδης για το Μεξικό. Εάν θέλουμε η Κανκούν να αποτελέσει μια επιτυχία, η χρηματοοικονομική αρχιτεκτονική των μηχανισμών που θα θεσπιστούν σε οικονομικό επίπεδο για να προωθηθούν οι δράσεις αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να τύχουν διαπραγματεύσει τουλάχιστον επί της αρχής. Θα πρέπει για να γίνει κάτι τέτοιο να υπάρξει οικοδόμηση εμπιστοσύνη μεταξύ όλων. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αναλυφθούν από τώρα ήδη δράσεις για την άμεση πρόσβαση των αναπτυσσομένων χωρών στα 30 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο που προβλέπεται να ξεκινήσουν από το 2010 μέχρι τα 100 δισεκατομμύρια που θα φτάσουν το 2020. Ελπίζουμε λοιπόν ότι με τον τρόπο αυτό δεν θα διαψεύσουμε τις προσδοκίες των χωρών αυτών και τις ελπίδες τους και θα δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εκταμείευση αυτών των κονδυλίων και εδώ ίσως υπάρχει ένα ψευδές δίλημα μεταξύ της κυριαρχικότητας και της εποπτείας το οποίο θα πρέπει να το ξεπεράσουμε. Όλες οι χώρες εξίσου έχουν μια ευθύνη και τόσο οι χρηματοδότε όσο και οι αποδέκτε θα πρέπει να παίξουμε το ρόλο μας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ελπίζω ότι έχω απαντήσει σε όλες τις ανησυχίες σας και τα ερωτήματά σας. Αλλιώς, κατά τα άλλα, είμαι πάντα στη διάθεσή σας στην Πρεσβεία του Μεξικού. Αν μέχρι την διάσκεψη Κανκούν έχετε κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα, αν θέλετε να έχετε περισσότερες πληροφορίες, προφανώς εξακολουθώ να είμαι στη διάθεσή σας και θα ήθελα πάρα πολύ να υπάρξει μια η αριθμητικά ισχυρή αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γεω Λάινεν και σας ευχαριστώ και πάλι για την ευκαιρία που μου δώσετε να λάβω το λόγο ενώπιον σας. ευχαριστώ πολύ κυρία Πρέσβη. Χαιρόμαστε και εμείς ιδιαίτερα για την έλευσή σας. Μας δώσατε ορισμένες νέες νοπές πληροφορίες. Προετοιμαζόμαστε για την Κανκούν την Τετάρτη θα κάνουμε μία βιντεοδιάσκεψη με την Κριστίνα Φιγγέρες, η οποία είναι διευθύντρια του, κλίματος, του τμήματος κλιματικής αλλαγής. Όπως σας είπα σε δύο εβδομάδες στο Στρασβούργο θα έχουμε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια θα μεταβεί μια αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διάσκεψη του Κανκούν. Νομίζω ότι θα είμαστε 33 βουλευτές. Αυτό δείχνει το πόσο θέλει να εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα είναι πολλοί άλλοι οι οποίοι θα μας συνοδεύσουν και εγώ εύχομαι και ελπίζω ότι η Μεξικανική Προεδρία θα είναι πράγματι επιτυχή γιατί αυτή τη στιγμή εσείς παίζετε το ρόλο μιας γέφυρας μεταξύ φτωχών και πλουσίων, μεταξύ βορρά και νότου και είναι σημαντικό το γεγονός ότι θέλετε να εξασφαλίσετε και την ε, διαφάνεια και τον περιεκτικό χαρακτήρα των διαπραγματεύσεων αυτών. Νομίζω ότι είναι πράγματι όλα αυτά μια εγγύηση ότι θα μπορέσουμε να έχουμε τις καλύτερες συνθήκες για να καταλήξουμε σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα και όλοι θέλουμε στο Μεξικό να έχουμε αυτή την επιτυχή κατάληξη. Λοιπόν, θα βρεθούμε και πάλι σε αυτή τη διαδικασία συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και μεγάλη και κάθε επιτυχία στο εγχείρημα αυτό της συνδιάσκεψης. Ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο της πρωινής μας συνεδρίασης. Την ε, πολλές φορές αναφερθήσα ήδη διάσκεψη βιοπικιλότητας στην, στην Αγκόγια. Ήταν 11 μέλη της, ε, τα μέλη της αντιπροσωπείας μας και κάποιους ε, από αυτούς τους βλέπω ήδη εδώ. Ο Επίτροπος Ποτότσνικ μας είχε ήδη ε, πληροφορήσει για όλα αυτά τα οποία θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Τα πράγματα λειτουργήσανε πολύ καλά. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και το έργο της Γραμματείας που μας βοήθησε να οργανώσουμε καλύτερα τις εργασίες μας και για μένα ήταν μια πολύ θετική έκπληξη για, το, για την ε, συνάντηση του δικτύου κλουμπ, του διακοινοβουλευτικού αυτού δικτύου που αντιμετώπισε όλα τα βασικά θέματα της βιοποικιλότητος και πιστεύω ότι το κλοπ θα πρέπει και στο μέλλον να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Είχαμε επίσης και ενημέρωση από μια σειρά χωρών, Νότια Αφρική, Ιαπωνία που ήταν ο αμφιτρίωνας της συνδιάσκεψης και επίσης συναντηθήκαμε και με την αντιπροσωπεία των Ηνωμένων Πολιτειών η οποία είχε χαρακτήρα μόνο παρατηρητού. Θα πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προσυπογράψει ακόμα αυτή τη σύμβαση για την βιοποικιλότητα και ίσως ήταν καλό ότι δεν ήταν παρόντες για αυτό το λόγο σαν συμμετέχοντες παρά μόνο ως παρατηρητές Βέβαια αυτό δεν τους έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις απόψεις τους και ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στην Κανκούν είναι φυσικά μέλη και όχι παρατηρητές, αλλά πάντα μια μεγάλη χώρα είναι καλό να βρίσκεται μέσα στην αίθουσα της διασκέψεως και όχι στους διαδρόμους. Είχαμε επίσης το Γενικό Γραμματέα της UNEP, τον Στάινερ, ο οποίος ε, ήταν παρόντες και ο οποίος μπορεί, ε, θα έρθει ευχαρίστως ενώπιον της Επιτροπής μας για να μιλήσει για την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση, την ε, διαδικασία του Ρίο, γιατί έχουμε τώρα πάρα πολλές συνδιασκέψεις, πάρα πολλές συμβάσεις, πάρα πολλά ταμεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί με τις διαδοχικές συνδιασκέψεις και ίσως θα πρέπει να τα σουλουπώσουμε όλα αυτά μέσα σε εισαγωγικά με την προοπτική της διάσκεψης του Ρίο το 2020. Ήταν επί ξηρού ακμής σε πολλές φορές η συνδιάσκεψη, δεν ήταν εγγυημένη η επιτυχία της, παρόλα αυτά μπορέσαμε να καταλήξουμε σε μια συνένεση στο τέλος. Όλα αυτά ήταν ε, δυνατόν να γίνουν μονάχα με αμοιβέ παραχώρησει και εμείς δεν μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε ότι όλα αυτά τα οποία είχαμε ζητήσει στο ψήφισμά μας, αλλά η COP10 μπόρεσαν να συμβάλλουν ιδιαίτερα να γίνει δεκτή η έννοια του φυσικού κεφαλαίου και των απολειών που έχουμε υποστεί στα πλαίσια του φυσικού κεφαλαίου στη γη μας, το γεγονός δηλαδή να, να διαπιστωθεί ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χάνουμε κάθε χρόνο φυσικούς πόρους και επομένως έχουν τεθεί ε, στρατηγική στόχη για το 2020, 20 τομείς από ό,τι διαπιστώσαμε. Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες, αλλά τουλάχιστον αυτό που επετέφθη στην Αγκόγια είναι ότι υπήρξε μια συνένεση σε αυτά τα θέματα. Το πρωτόκολλο ABS επίσης ήταν και αυτό αντικείμενο συζητήσεων στην ε, Αγκόγια. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια ισοδίκαια κατανοή των πόρων μεταξύ των λαών που πρέπει να τους χρησιμοποιήσουν για την επιβίωσή τους. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αμερικανικές εταιρείες οι οποίες δεν δεσμεύονται από αυτή τη συμφωνία και αυτό οδηγεί σε μια στρέβλωση και του ανταγωνισμού. Ίσως το πιο αδύνατο σημείο της Ναγκόγια ήταν το θέμα της κινητοποίησης χρηματοοικονομικών πόρων. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπόρεσε να προχωρήσει ακόμα και αυτή σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις. <clears throat> Και φυσικά το γεγονός ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν απούσες έφερε στο επίκεντρο της προσοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά ήταν στο κέντρο και των διαπραγματεύσεων και των συμβιβασμών που επιτέθησαν στο τέλος και εγώ θέλω να επενέσω την Κομισιόν για το έργο της <clears throat> και για το γεγονός ότι μπόρεσαμε να μιλάμε με μία μονάχα φωνή και αυτό φυσικά ήταν και αποτέλεσμα των προσπαθειών της Βελγικής Προεδρίας για να μπορέσει να προωθηθεί περαιτέρω το πρωτόκολλο ABS <clears throat> περισσότερο να διευρυνθεί και να είναι πολύ πιο ε, πλήρες από ό,τι στην ε, έναρξη της ε, συνδιάσκεψης της Ναγκόια και η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πράγματι κάτι το οποίο ήταν υποδειγματικό για να μπορέσουν να εξευρεθούν <clears throat> συμβαστικές λύσεις και με άλλες ομάδες χωρών και ιδιαίτερα με τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αυτά λοιπόν υπομορφήν εναρκτήριων παρουσιάσεων και θα δώσω ευχαρίστως το λόγο σε όλους αυτούς οι οποίοι θέλουν να πούν κάτι. Ευχαριστώ Πρόεδρε, δεν πρόκειται να επαναλάβω αυτά τα οποία είπατε και εγώ συμμερίζομαι τα αισθήματά σας όσον αφορά την αντιπροσωπεία μας. Λίγο, λίγα λόγια, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν είναι πλήρες μέλος της σύμβασης. Ίσως ε, αυτό να, ήταν, να είχε και θετικές πτυχές, διότι πιστεύω ότι ε, οι, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα είχαν ποτέ συμφωνήσει με αυτό το πρωτόκολλο του μοιράσματο αν θέλετε, των ε, κερδών των πλεονεκτημάτων, λόγω ακριβώς των, της πίεσης ε, της φαρμακο, φαρμακευτικής βιομηχανίας τους, όμως με ανησυχεί λίγο η όλη διαδικασία επικύρωσης της σύμβασης, γιατί πιστεύω ότι κάποια από τα κράτη-μέλη και κάποιες κυβερνήσεις, κάποια κοινοβούλια θα το ξανασκεφτούν το θέμα, κυρίως και ίσως αλλάξουν άποψη, κυρίως αν αφορά το πρωτόκολλο για την πρόσβαση και τον κατανομή, αν θέλετε, των πλεονεκτημάτων. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσουν τελικά. Τώρα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την, και ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο για τον ανοιχτό τρόπο και ε, με τον οποίο μας ενημέρωναν κάθε βράδυ. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να εξελιχθεί μια τέτοια συνεργασία. Θα ήθελα και εδώ να του ευχαριστήσω επίσημα. Ε, κάτι με απογοήτευσε όμως. Ήλπιζα πριν από τη σύμβαση ότι θα υπήρξε μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κόσμου για τη σημασία της βιοπικιλότητας, λαμβάνοντας υπόψη τον περιορισμένο ενδιαφέρον του τύπου, πιστεύω ότι αυτός ο στόχος δεν επιτεύχθηκε. Αυτό επομένως είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να δουλέψουμε παραπάνω. Ένας τρόπος για να γίνει κάτι τέτοιο είναι να περιορίσουμε το χάσμα ανάμεσα στην περιβαλλοντική βιοπικιλότητα και την οικονομική πτυχή του θέματος. Ε, επομένως, Πρόεδρε, μήπως θα μπορούσαμε να έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων εδώ στο Κοινοβούλιο για να συζητήσουμε την διεπικελότητα όχι μόνο από την περιβαλλοντική πτυχή αλλά και από την οικονομική πτυχή. Ίσως θα μπορούσαμε να καλέσουμε τον κύριο Πάβα Σούμφενκ για να μας πει όχι μόνο ε, τι πρεσβεύουμε, για να ακούσουμε μάλλον, να συζητήσουμε όχι μόνο τι πρεσβεύουμε εμείς, αλλά και τι πρεσβεύουν οι συνάδελφοι από την Οικονομική Επιτροπή. Όλος έγινε ένα θέμα για, το πρωτόκολλο και συζητήθηκε το πρωτόκολλο αυτό και, στο, και στην Αγκόγια και τα θέματα ευθύνη και τα, η οικονομική η οικονομία μάλλον του, των φυσικών πόρων, των, των περιβαλλοντικών πόρων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Η Σαντρίν Μπελιέ. Ευχαριστώ. Και εγώ να μην ξαναπαναλάβω τους αυτά που είπαν οι προαλληλήσαντες. Ε, ήθελα να υπογραμμίσω την, την ποιότητα της οργάνωσης, ε, τη δουλειά που έκανε η Γραμματεία της Επιτροπής για το Περιβάλλον. Ε, πρέπει να το μόνο σε αυτό. Επίσης, να ευχαριστήσω τη συνεργασία που είχα και ήταν πλούσια και μας επέτρεψε σαν Ευρωπαίοι βουλευτές να μπορέσουμε να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε σωστά στα πλαίσια αυτής της ενεργασίας. Είχαμε και την Προεδρία του Συμβουλίου. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες εργασίας ήταν ιδανικές θα έλεγα. Επίσης να ευχαριστήσω γιατί ανακάλυψα εγώ στο, το ρόλο που μπορούσε να παίξει κανείς το ρόλο της βιοποικιλότητας και σε άλλους ε, τομείς για το περιβάλλον. Και το θέμα ότι είχα μια σωστή εργασία και συνεργασία με το Είχε δημιουργηθεί ένα πολύ καλό περιβάλλον εμπιστοσύνης εκεί στην Αγκόγια, κάτι που μας επέτρεψε να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. οι τρεις συμφωνίες υπογράφησαν ε, μια μισή το πρωί. Πετύχαμε δηλαδή μια συμφωνία. Και όσον αφορά από εμά, πέρα από τις φιλοδοξίες που είχαμε, ε, έχουμε μια ικανοποίηση διότι ε, δημιουργούνται ελπίδες σε ένα άλλο επίπεδο και συνεργασίες πολυμερείς για μια νέα διακυβέρνηση όσον αφορά το μέλλον στα πλαίσια του περιβάλλοντος. Επίσης, ένα πολύ καλό νέο όσον αφορά τη βιοπικιλότητα, διότι αυτό θα μας επιτρέψει να περάσουμε ε, σε, καλύτερες, ε, σε καλύτερες, ε, καλύτερο αποτέλεσμα από το Κιώτο Επίσης να πω ότι έχουμε και ένα άλλο καλό νέο όσον αφορά την οικοδόμηση συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για στα πλαίσια της συνθήκες μετά τη Λισαβόνα για να μπορέσουμε από τώρα μέχρι το μέλλον να πάρουμε μια θέση να προσδιοριστούμε στα πλαίσια της, ε, ενός παγκοσμίου επίπεδου σαν μια δύναμη και πιστεύω ότι κάτι ακόμα που ήταν θετικό σε αυτές τις διαπραγματεύσεις είναι ότι βλέπουμε μια νέα δύναμη σε, αυτό, σε αυτή τη σκακέρα θα λέγαμε σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ξέρουμε εμείς, το είπε και η Επιτροπή, εμείς εδώ σε αυτήν εδώ την Επιτροπή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βλέπουμε τη στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία συζητείται για την περίοδο 2011-2016 βλέπουμε τι διακυβεύεται και πραγματικά ελπίζουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να κρατήσει τον ηγετικό της ρόλο σε αυτά τα πλαίσια. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια γιατί μείνατε μέχρι το τέλος. Πραγματικά Ε, ήταν δύσκολες εμπραγματεύσεις και πραγματικά και δεν είναι ε, χρήσιμο να απομακρύνεται κανείς από τις διαπραγματεύσεις ε, τη στιγμή που γίνονται θα πρέπει κανείς να πάει μέχρι το τέρμα και ξανά σας συγχαίρω γι' αυτό. Η Κάριν Κάλεμπαχ. Και εγώ θα δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μην ευχαριστήσω όλους για την διοργάνωση της ε, διάσκεψης και συμφωνώ με τη Σαντρίν. Θα ήθελα να τονίσω όμως κάτι ακόμα, το οποίο αναφέρθηκε από ένα προαναλύσαντα συνάδελφο. Νομίζω ότι ένας αποφασιστικός παράγοντας στην επιτυχία της συνδιάσκεψης ήταν το γεγονός ότι και στα πλαίσια της μελέτης TIP είχε τονιστεί η σημασία που έχουν τα λειτουργούντα οικοσυστήματα και πώς μπορεί να αξιολογήσει κανείς τα οικοσυστήματα αυτά και ότι όλα αυτά δεν είναι μοναχά στο μυαλό ορισμένων επιστημόνων, δεν είναι σενάρια τρόμου ότι θα χάσουμε ζωικά και φυτικά είδη και θα χάσουμε βιοπικιλότητα, αλλά ότι αντίθετα όλα αυτά μπορούν να είναι καταμετρήσιμα και να αντιμετωπιστούν σε συγκεκριμένα σχέδια. Και φάνηκε επίσης ε, αυτό και στις συνεντεύξεις τύπου στη χώρα μου πολλές φορές ε, νομίζουν οι δημοσιογράφοι ότι όλα αυτά τα κάνουμε για να προστατεύσουμε τις ορχιδέες ή κάποιους βατράχους ή κάτι τέτοιο. Είναι πολύ περισσότερα αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Δεν είναι μονάχα συγκεκριμένα και μονάχα είδη που θέλουμε. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε την επιβίωση ενός συνολικού συστήματος και γι' αυτό κάνω αυτή την έκκληση προς όλους τους συναδέλφους να κατανοήσουμε ότι πρέπει να μπορέσουμε και στα ίδια μας τα κράτη-μέλη να λειτουργήσει η προστασία της βιοποικιλότητας και επίσης και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε και περισσότερα πράγματα και στις χώρες μας. Ο, φόρος μου, φόβος μου βέβαια είναι ότι δεν θα προχωρήσει το θέμα της χρηματοδότησης της βιοποικιλότητας. Όπως ελέγχθη, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν συμμετέχουν στη Σύμβαση Βιοποικιλότητας. Οι άλλοι οι οποίοι συμμετέχουν στη διάσκεψη αυτήν, κυρίως αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίοι θα είναι αποδέκτες κονδυλίων, θα πρέπει εμείς να έχουμε λοιπόν επίγνωση ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει ένα κομμάτι, ένα μεγάλο κομμάτι του χρηματοδοτικού βάρους και αυτό σημαίνει ότι και στα κράτη-μέλη μας θα πρέπει να ενσωματωθεί η προστασία της βιοποικιλότητας σε όλες τις πολιτικές των ε, κρατών μελών μας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό σημαίνει πράγματι όπως ελέγχει περισσότερη συνεργασία με τους συναδέλφους από την Οικονομική Επιτροπή. Η Άννα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Όπως και η προλαλήσασα, θεωρώ ότι είχαμε μια συμφωνία της τελευταίας στιγμής και συγχαίρω και εγώ πάλι τη συναδέλφισσα που έμεινε μέχρι το τέλος. Υπάρχουν όμως κάποια πράγματα που με ενοχλούν. Ήταν καλό να έχουμε μια τέτοια σειρά ε, καλών συμφωνιών σε υψηλό επίπεδο, αλλά τι θα αλλάξει με αυτό όσον αφορά τα είδη τα οποία απειλούνται. Τι θα γίνει ε, ή κάποια άλλα είδη τα οποία απειλούνται στη θάλασσα, στα δίκτυα των ψαράδων. Ε, προβλήματα που δημιουργούνται με τις πολυεθνικές εταιρείε. Μήπως είναι πιο υπεύθυνε όσον αφορά ε, το θέμα του... της ασφάλειας. Είναι σημαντικό να μπορέσουμε να ελέγχουμε εμείς ε, και να το δούμε νομοθετικά και θα ήταν καλό που που το βλέπω σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να δούμε Έχουμε δρόμο να διανύσουμε σε σχέση δηλαδή με την Αφρική, την Κίνα και τη Λατινική Αμερική. Πραγματικά υπάρχουν πολύ μεγάλες προκλήσεις για να μπορέσουμε να περάσουμε στην εφαρμογή όλων αυτών εδώ των μέτρων. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς, θα ήθελα να συγχαρώ την αντιπροσωπεία, ειλικρινά. Έκαναν πολύ καλά τη δουλειά τους, γιατί τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. Η φιλοξενούσα χώρα, η Ιαπωνία, έκανε την αλλαγή. Να μας, πει, να μας πείτε κι εσείς και η Σαντρίν πιο συγκεκριμένα που έμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή. Ποια ήταν η προστιθέμενη αξία της Ιαπωνίας πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τις φιλοξενούσες χώρες ε, να βελτιώσουν τις παροχές τους. Επίσης για το ABS, ποιος ήταν ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρνητικός ρόλος τελικά στις διαπραγματεύσεις στην Αγκόγια. Για το ABS, ποιος... και συμφωνώ με τα σχόλια που έκανε ο Άικχαρτ και η Σάτου Χάση για το πώς μπορεί να βελτιωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύσει στο Γανκούν. Επίσης, θα πρέπει να βελτιώσουμε τις θέσεις μας στις διαπραγματεύσεις, γιατί από ό,τι φαίνεται ότι σε πολλά σημεία πρέπει να βελτιωθούμε. Έστω και αν σε γενικές γραμμές είμαστε στη σωστή πορεία. Υπάρχουν όμω περιθώρια βελτίωσης και σε σημεία που είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Ευχαριστώ. Τελευταίος ομιλητής κ. Σέρκα. Κοιτάξτε, θα ήθελα να ευχαριστήσω την Γραμματεία γιατί οργάνωσε την όλη συνάντηση. Θα πρέπει να ευχαριστήσουμε την Παραονζάρ και το Γιώστα για, για τη βοήθειά τους. Μία ερώτηση, μία διαδικαστική για μία επί του περιεχομένου. Αυτή η συνάντηση στην Αγώγια έδειξε ότι η Ευρώπη μπορεί να μιλήσει με μία φωνή και το έκανε γιατί ακριβώς υπήρξε πάρα πολύ καλή συνεργασία ανάμεσα στην Βελγική Προεδρία και στην Επιτροπή. Και αυτό είναι σημαντικό και κρίσιμο στα επόμενα βήματα προς το Κανκούν, διότι η Κομισιόν ε, μιλούσε για το IBS, ε, Access and Benefit Sharing, και ο Επίτροπος Ποτάτσνικ και, η Επιτροπή και τα μέλη της Επιτροπής ε, Περιβάλλοντος ε, μπόρεσαν να μιλήσουν ε, με μία φωνή ενώ σε άλλα θέματα ήταν η Βελγική Προεδρία που είχε το πρώτο ρόλο. Άρα αυτή η κατανομή των αρμοδιοτήτων ήταν πάρα πολύ χρήσιμη και δεν θα πρέπει να βλέπουμε και τα θέματα τελείως σφαιρικά. Πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο γιατί και εκεί και αυτό θα πρέπει να γίνει και στο Κανκούν. Αρκεί να είναι ένα ο υπεύθυνο βέβαια. Τώρα, εν συντομία, Πρόεδρε, για το μπορούμε να είμαστε ευχαριστημένοι με τα αποτελέσματα. Μεν, το πρόβλημα είναι η εφαρμογή. Μπορούμε να συμφωνήσουμε για τους στόχους, ε, για να αποφασίσουμε για άλλα πράγματα. Αλλά οι στόχοι αυτοί σημαίνουν κάτι. Το να μειώσουμε τις επιβλαβείς ουσίες για την βιοπικιλότητα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα οικοσυστήματα. Και αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί και πρακτικά στις εσωτερικές μας πολιτικές. Αυτό είναι το θέμα. Εάν αρχίσουμε να συζητάμε για την γεωργική μεταρρύθμιση, Προφανώς, αν ε, μιλάμε για την φθήνουσα πορεία των ε, επιβλαβών ε, ουσιών, θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας στην γεωργική μεταρρύθμιση. Θα πρέπει οι συνάδελφοι που ασχολούνται με αυτούς και που θα πρέπει να εφαρμόσουν με αυτούς τους στόχους, θα πρέπει να τους εφαρμόσουν στην γεωργική μεταρρύθμιση, ουσιαστικά πλέον. Τώρα για την Ιαπωνία εφόσον μιλάμε για εθνική, όταν αρχίσουμε να μιλάμε για εθνική βιοπικιλότητα και εθνική προστασία, είμαστε πολύ φιλόδοξοι και αυτό ακριβώς κάνει η Ιαπωνία. Έχουν πολύ φιλόδοξες πολιτικές και πολύ φιλόδοξου στόχου για την βιοπικιλότητα. Απ' την άλλη πλευρά όμω, αυτό το οποίο κάνουν με την αλία εκτό των χωρικών υδάτων τη Ιαπωνία είναι μια άλλη ιστορία. Επομένω, θα πρέπει να υπάρχει μια συνέπεια ανάμεσα στα οποία ε, ε, εφαρμόζουμε στο εσωτερικό τη χώρα μα και αυτά τα οποία κάνουμε στο εξωτερικό τη χώρα μα. Και εκεί η Ιαπωνία έχει περιθώριο βελτίωση. Και η Ευρώπη βέβαια έχει ε, περιθώριο βελτίωση. Επομένως θα πρέπει τους στόχους για τους οποίους δώσαμε μάχη στην Αγκόλια να τους λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Αυτά λέει ο πρόεδρος, ευχαριστώ. Νομίζω ότι η Ιαπωνία είναι η μόνη η οποία έβαλε και χρήματα στο τραπέζι, 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά προσέφερε η φιλοξενούσα χώρα. Βοήθησε να έχουμε μια καλύτερη ε, ατμόσφαιρα και μετά διευκόλυναν και την ε, συνεδρίαση με διαφόρους ε, διαμεσολαβητές για τον Βορρά και για τον Νότο και το ίδιο η εφάρμοση και για την χρηματοδότηση και γιατί ούτω ή άλλω δεν μπορούμε να έχουμε μια γενική συζήτηση με όλε τι συμμετέχουσες χώρε. θα πρέπει να δημιουργηθούν διάφοροι πυρήνε. Και αυτό είναι ένα χρήσιμο δίδαγμα και για το Κανκούν. Επίση, θα πρέπει να, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα με την επικύρωση των, του πρωτοκόλου και στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και το mainstreaming αν θέλετε τη βιοπικιλότητας και στις άλλε πολιτικέ. Θα πρέπει να εντάξουμε τη βιοπικιλότητα και στι διάφορε. Ε, πολιτικές ε, τις κοινοτικές. Θα πρέπει μετά τον Γενάρη να δούμε τι έγινε, όπου ο Επίτροπος θα πρέπει να έρθει να μας ενημερώσει γιατί γίνεται με την διοπικιλότητα και στις άλλες πολιτικές. Το Globe τώρα ε, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τους νομοθέτες. Θα πρέπει να κάνουμε ανταλλαγές με διάφορες χώρες και να συμμεριστούμε τις εμπειρίες μας ε, με τις χώρες αυτές που θέλουν να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό. Αυτή ήταν η Ναγκόγια, με λίγα λόγια. Και ελπίζουμε ότι και η ανθρωπότητα και τα Ηνωμένα Έθνη πιο συγκεκριμένα θα μπορέσουν να καταλήξουν μια συμφωνία. Ας δούμε τι θα γίνει στην επόμενη διάσκεψη στο Κανκούν. Τελείωσε εδώ η πρωινή μας συνεδρίαση και θα ξαναβρεθούμε στις 3 η ώρα με τον πρόεδρο της ΕΤΣΑ. Του ΕΤΣΑ μάλλον. Δεν έδωσε τον ρόλο στην Κομισιόν, αλλά θα καλέσουμε